Αγαπητοί μου φίλοι της Επιτροπής Ήτρε, σας είμαι ευγνώμων που ε, ήρθατε. Εμείς οι τέσσερις τουλάχιστον. Πολύ μεγάλος αριθμός. Αλλά είμαι βέβαιος ότι σε λίγα λεπτά θα καταφτάσουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Ας περιμένουμε λοιπόν ακόμη δύο-τρία λεπτά για τους υπόλοιπους. <clears throat> Καλημέρα σας και πάλι και καλώς ήρθατε στην τρίτη φάση της συνεδρίασης της Επιτροπής Ήτρε. Το πρώτο θέμα είναι η ανταλλαγή απόψεων για την εφαρμογή του πρίμα και τη σύναψη διεθνών συμφωνιών. Όπως γνωρίζουμε το θέμα είναι σημαντικό γιατί το πρίμα είναι μια σύμπραξη μεταξύ φορέων δημοσίου με συμμετοχή και τρίτων χωρών. Οπότε είναι κάπως πιο περίπλοκο από το να συμμετέχουν μόνο ε, κοινωτικέ χώρες. Και μάλιστα στο μέλλον κάποιες χώρες που δεν συμμετέχουν ε, ήδη στο πρόγραμμα Horizon 2020 πρέπει να διαπραγματευτούν μια επιστημονική και τεχνολογική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να μπορέσουν να λάβουν μέρος στο πρίμα. Τέσσερις από τις διαπραγματεύσεις αυτές έχουν ήδη διεκπαιρεωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Αλγερία, Αίγυπτο, η και Λίβανο, τέσσερις χώρες δηλαδή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει τη συνένεσή του, τη συγκατάθεσή του για αυτές τις συμφωνίες προκειμένου να τεθούν σε ισχύ. Και μάλιστα το πρίμα έχει προγραμματιστεί να λειτουργήσει από τον Ιανουάριο του 2018. Οπότε βιαζόμαστε γιατί ούτε ένα τρίμηνο δεν μας έχει μείνει. Η κυρία Σακοράφα είναι η συγγητριά μας για το θέμα το πρίμα, οπότε παρακαλώ κυρία Σακοράφα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την νέα εταιρική σχέση στον τομέα της έρευνας και της κοινωνία στην περιοχή της Εμεσογείου Πρίμα τον περασμένο Ιούλιο με συντριπτική πλειοψηφία. Πρόκειται για την πρώτη εταιρική σχέση με νομική βάση το άρθρο 185 της Συνθήκης που αφορά στις συμπράξεις μεταξύ δημοσίων φορέων και επικεντρώνεται στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή αυτή της Μεσογείου, περιλαμβάνοντας τη συμμετοχή γειτονικών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με δεκαετή ορίζοντα υλοποίηση και έναρξη εφαρμογή την 1η Πρώτου του 2018, ο γενικό σκοπό του πρίμα είναι η ανάπτυξη και η υιοθέτηση καινοτόμων και ολοκληρωμένων λύσεων για τη βελτίωση τη απόδοση, της ασφάλειας, της προστασίας και της βιωσιμότητας των συστημάτων γεωργικών προϊόντων διατροφής και της παροχής και διαχείρισης των υδάτων της περιοχής της Μεσογείου. Ο γενικότερος στόχος του πρίμα είναι να συμβάλλει στη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη στο πλαίσιο της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης ενώ ο ειδικό του στόχο αφορά στον συντονισμό και την ενίσχυση των εθνικών προγραμμάτων έρευνα και καινοτομία στου τομεί που πραγματεύεται, στο πλαίσιο μια πολυπαραγωγική, πολυδιάστατη και ολοκληρωμένη προσέγγιση. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι ένοπλε συγκρούσει, οι εξωτερικέ επεμβάσει, οι διώξει, οι εθνοτικέ καρθάρσει, η γενικευμένη βία, η πολιτική αστάθεια, ο θρησκευτικό φονταμενταλισμό, η αλλαγή του κλίματο, οι φυσικέ καταστροφέ, η μη βιώσιμη διαχείριση των πόρων και η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού αναδεικνύονται σαν πιο κρίσιμοι παράγοντε που συμβάλλουν στον αναγκαστικό εκπαρτισμό και στη μετανάστευση. Αυτό το φαινόμενο έχει εξελιχθεί σε μια τεραστίου μεγέθου ανθρωπιστική κρίση, μια κρίση που είναι ωστόσο το φυσικό αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών και παρεμβάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η προσέγγιση του πρίμα και συγκεκριμένα η αναζήτηση αφενός βραχυπρόθεσμων λύσεων για την άμεση αντιμετώπιση της μεταναστευτικής πίεσης και φετέρου σημαντικών δομικών επενδύσεων για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης και του αναγκαστικού εκπατρισμού αποτελεί μια πρωτοβουλία που κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Αγαπητοί συνάδελφοι, Όπω έχω τονίσει κατά επανάληψη με την ιδιότητα τη εισηγήτρια τη βασική πράξη, θεωρώ το πρίμα μια σπάνια προσπάθεια επιστημονική διπλωματία τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέχρι στιγμή η σημαντικότερη ευρωμεσογειακή πρωτοβουλία στον τομέα τη έρευνα και τη καινοτομία, μια μοναδική ευκαιρία για τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τι τρίτε χώρε τη Μεσογείου να ενώσουν τι δυνάμει του και αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα για το πώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι πραγματικά ανοιχτή για συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο. 19 συνολικά χώρε μετρέχουν από κοινού στο πρίμα. 11 κράτη-μέλη, 3 συνδεδεμένε χώρε με το πρόγραμμα Ορίζοντα 2020 και πέντε τρίτε χώρε με τι οποίε και όπω ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφο 2 τη σχετική απόφαση θα πρέπει να συναυθούν συμφωνίε διεθνή, επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία. Ω εκ τούτου, μετά την έγκραση του πρίμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύτηκε μια σειρά από διεθνεί συμφωνίε με τι εν λόγω τρίτε χώρε. Καλωσορίζω λοιπόν στο σημείο αυτό την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις συμφωνίες επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας με την Αλγερία, την Αίγυπτο, την Ιορδανία και το Λίβανο, η διαπραγμάτευση των οποίων έχει ήδη ολοκληρωθεί και καλώ όλα τα μέλη της ΣΥΤΡΕ να παράσχουν τη συγκατάθεσή τους στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας, ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή των εν χωρών στο πρίμα από την έναρξη εφαρμογής του τον Ιανουάριο του 2018. Thank Σας ευχαριστούμε. Και τώρα θα δώσω το λόγο στους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Εκ μέρους του ΕΛΚΟ, κύριος Ρούμπιχ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίζω αυτή την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Για, για μας είναι σημαντικό να βελτιωθεί η επιστημονική εργασία και νομίζω ότι στι χώρε αυτέ υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία να δραστηριοποιηθούμε. Αν τεθούν όλα αυτά λοιπόν σε ίσχυ το 2018, θεωρώ ότι θα υπάρξει μεγάλο πλεονέκτημα. Και επίση θα ήθελα να υπογραμμίσω το εξή. Σε ό,τι αφορά την Ιορδανία, είναι καλέ οι επαφέ. και θα έχουμε και το σχετικό φόρουμ που θα διοργανωθεί. Νομίζω ότι το φόρουμ αυτό λοιπόν θα μπορούσε να αποτελέσει μια πλατφόρμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να ενισχυθεί η επιστημονική συνεργασία. Συμμετείχαμε και στο φόρουμ STS στην Ιαπωνία και αυτό είναι εξωσημείωτο. Συμμετείχαν βραβευμένοι με το βραβείο Νόμπελ που συζήτησαν παγκόσμια προβλήματα και σε ό,τι αφορά τις συζητήσεις, μπήκαν στον επίκεντρο οι στόχοι της χιλιετίας. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να μπουν στον επίκεντρο αυτοί οι βιώσιμοι στόχοι και η Επιτροπή Ήτρε λοιπόν κατεξοχήν θα πρέπει να θέσει νέες προτεραιότητες για να τονίσει τον κλάδο της ενέργειας, φυσικά την έρευνα και την, την ανάπτυξη. Γι' αυτό λοιπόν η συνεργασία με τις χώρες αυτές είναι ιδιαίτερως σημαντική. 17 Μαΐου του χρόνου θα προσπαθήσουμε και με το φόρουμ STS να ενισχύσουμε ακριβώς την ε, διεθνή αυτή πλατφόρμα και γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι το πρόγραμμα αυτό είναι κέρια σημασία για μας και θα το υποστηρίξουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και Πρόεδρος. Εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών η κυρία Καβεσόν Ρουίς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να εκφράσω την ικανοποίησή μου, γιατί βλέπω ότι το πρίμα ακολουθεί την πορεία του και θα ήθελα να γνωρίσω την προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέρ του πρίμα προκειμένου να προωθηθεί, δρομολογηθεί αυτό το πρόγραμμα και επίσης εγκρίθηκε πρόσφατα τον Ιούλιο. Εκφράζω μεγάλη ικανοποίηση για τις εξελίξεις αυτές. Επίσης χαίρομαι για τις διεθνείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τρίτες χώρες όπως Αλγερία, Αίγυπτος, Ιορδανία και Λίβανο και ε, θεωρώ ότι τα πράγματα είναι πολύ ικανοποιητικά. Ε, 11 είναι οι ευρωπαϊκές χώρες, 8 από τη Μεσογειακή Λεκάνη και θα προσπαθήσουν να βρουν λύσεις στα 180 εκατομμύρια κατοίκους της περιοχής της Μεσογείου που αντιμετωπίζουν προβλήματα είτε με τη διαχείριση δάτινων πόρων είτε ως προς την επιστημιστική τους ασφάλεια. Και νομίζω ότι θα είναι υπόδειγμα διπλωματικής, ε, επιστημονικής διπλωματίας που θα συνάδει υπέρ της ανάπτυξης και της βιώσιμης διαχείρισης. Και μάλιστα η χρηματοδότηση εξασφαλίζεται στο ένα τμήμα της από τον ορίζοντα 2020 και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε παρόμοια σχέδια και προγράμματα. Αυτά προς το παρόν. Περιμένουμε τακτική ενημέρωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πορεία εφαρμογής ε, του προγράμματος Πρίμα και θα συμβάλλω όσο μπορώ για να στεφθεί με επιτυχία σε όλες τις φάσεις αυτό το πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το πρόγραμμα Πρίμα πραγματικά παρουσιάζει αρκετά ενδιαφέροντα σημεία. Εμείς ε, έχουμε τοποθετηθεί επί της αρχής όταν συζητήσαμε το πρίμα και κατά πόσο θα έπρεπε να εγκριθεί. Είχαμε ε, υποβάλει αρκετές σκέψεις και ενστάσεις γύρω από τα προβλήματα τα οποία παρουσιαζόταν. Σε σχέση με το σκοπό πρώτα απ' όλα θεωρούμε βεβαίως ότι είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα. <clears throat> πρέπει να ενισχύσουμε την επιστημονική διπλωματία, πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες στο θέμα της ε, ενέργειας, στο θέμα της έρευνας και της τεχνολογίας, στη διαχείριση των ε, υδάτων ως εκ τούτου, οι στόχοι αυτοί βεβαίως μπορούν να συμβάλλουν στο να μειωθούν ε, οι μεταναστευτικές πιέσεις ε, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι οι πόλεμοι, η φτώχεια αλλά και η κλιματική αλλαγή δημιουργούν ε, τεράστιες μεταναστευτικές πιέσεις. Από εκεί πέρα βέβαια θέλουμε να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα <clears throat> θεωρούμε ότι όλη η προσπάθεια εντάσσεται σε αυτό που ονομάζουμε μεταβλητή γεωμετρία διότι βλέπουμε να συμμετέχουν μόνο 11 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε ένα στόχο ο οποίος αφορά όλους. Διότι το να μειωθούν οι μεταναστευτικές πιέσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αφορά την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, τις χώρες του Νότου. Αφορά όλη την Ευρώπη. Επομένως, ε, πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχει συνολική συμμετοχή των κρατών μελών. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι παρακολουθούμε ένα ιδιαίτερα ενισχυμένο ρόλο που αποδίδεται στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ε, για τις οποίες έχουμε πάρα πολλά ερωτηματικά ως προς τον τρόπο διαχείρισης αναπτυξιακών έργων και στις τρίτες χώρες, ε, αλλά και στην ε, ίδια την Ελλάδα και την Ιταλία, στη διαχείριση κονδυλίων για τις μεταναστευτικές ροές. Έχουμε καταγγείλει επανειλημμένα ότι γίνεται πάρτι από διάφορες ΜΚΟ που αξιοποιούν τα κονδύλια τα οποία είναι για τους πρόσφυγες, για τους μετανάστες. Στο τέλος δεν φτάνουν αυτά τα αποτελέσματα υπέρ των ίδιων των προσφύγων και των μεταναστών. I'm going to finish, Mr. Chairman, in one minute. Ε, ε και επίσης ε, έχουμε υποβάλει και ιδιαίτερε ενστάσεις για τη συμμετοχή της Τουρκίας η οποία επί του πρακτέου όχι μόνο δεν διευκολύνει τα, τα ζητήματα ε, για τα οποία έχει συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά έχει γεμίσει πλέον τα νησιά του Αιγαίου με πολλούς πλέον πρόσφυγες και κυρίω παράνομου μετανάστε. Αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστιο πρόβλημα στα νησιά του Αιγαίου. Εν πάση περιπτώσει εμείς ε, θα σταθούμε θετικά σε όλη αυτή την προσπάθεια, θα, είμαστε, ε, θα συμμετέχουμε. Θέλουμε να λάβουμε γνώση αναλυτικά των διεθνών συμβάσεων που έγινε με Αλγερία, έγιναν με Αλγερία, Αίγυπτο, Ιορδανία και Λίβανο, να δούμε το περιεχόμενο. Πιστεύουμε ότι πρέπει να ενημερώνεται τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και φυσικά θα συμμετέχουμε με παρεμβάσεις και τροπολογίες στην όλη διαδικασία την οποία από ό,τι βλέπω πρέπει να έχουμε τελειώσει μέχρι το τέλος του χρόνου διότι είναι πλέον μια ευσπεσμένη διαδικασία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you much, συνάδελφοι. Από τους φιλελεύθερους, εκπρόσωπος. Εκ μέρους του κυρίου Τελίτσκα. Υποστηρίζω την εταιρική αυτή σχέση για την έρευνα και την κοινοτομία στον χώρο της Μεσογείου, το λεγόμενο πρίμα. Και το υποστήριξα από την αρχή. Δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να προωθήσει την κοινοτομία στον τομέα της γεωργίας, των διατροφικών συστημάτων ή διαχείρισης του νερού, είναι και ένα εργαλείο επιστημονικής διπλωματίας, όπως είπε και η συγγήτρια. Αν επιτρέψουμε σε αυτό το πρόγραμμα να αναπτυχθεί θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής, θα βρεθούν λύσεις σε πιεστικά προβλήματα προσαρμογής ε, στο, στην κλιματική αλλαγή και μετριασμού των επιπτώσεων, αλλά θα διευκολυνθεί και ο διάλογος ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις τρίτες χώρες Μεσογείου. Τον Ιούλιο του 2017 συμφωνήσαμε με το Συμβούλιο και την Κομισιόν για το τελικό κείμενο της πρότασης. Ως κοιόδηση συγγήτρια για αυτό το θέμα, ε, ο Πάβελ πιστεύει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος το πρόγραμμα αυτό να μην ξεκινήσει. Και καλό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει τη συνένεσή του στα όσα έχουμε συμφωνήσει με την Αίγυπτο, ε, η Ορδανία, Λίβανο και Αλγερία. Δεδομένη τη τεράστια σημασία και, ε, και στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια, πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υποστηρίξει το πρόγραμμα αυτό. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Από τους πράσινου. Ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι μια μεγάλη πρωτοβουλία και πρέπει να ευχαριστήσουμε και την Κομισιόν αλλά και το Κοινοβούλιο για την γρήγορη εξέταση. Σε όλες τις μελέτες βλέπουμε ότι η κλιματική αλλαγή θα δημιουργήσει πρόβλημα στα δάση, στη γεωργία, στο πόσιμο νερό στις χώρες αυτές. Επομένως, έχουμε κάθε συμφέρον να πιέσουμε να προχωρήσει αυτή η επιστημονική συνεργασία γρήγορα και σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό θα πρέπει να γίνει χωρίς να πολιτικοποιήσουμε πάρα πολύ αυτό το φάκελο. Ε, δυστυχώς, ε, κύριε Μαριά, δεν συμφωνώ μαζί σας μαζί σας ότι θα πρέπει να τα ανακατέψουμε αυτά τα θέματα με τις ΜΚΟ και με την μετανάστευση. Θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι όταν σώζουμε ζωές στη Μεσόγειο και όταν έστω και μια ζωή δεν πεθαίνει από πνιγμό στη Μεσόγειο. Η κυρία Γιούσο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι υπόθηκαν όλα. Όπω είπε και ο τελευταίο ομιλητή, το θέμα αυτό είναι άσχετο με την ε, μετανάστευση. Είναι επιστημονικό θέμα που αφορά το περιβάλλον κυρίω. Η σημασία του πρίμα είναι τεράστια. Και γιατί έχουμε εδώ πέρα συγκεντρωθεί, γιατί συνεδριάζουμε, γιατί χώρε τρίτες χώρες που δεν ανήκουν και δεν συμμετέχουν στον ορίζοντα 2020, με βάση το άρθρο 1, παράγραφος 2, θα πρέπει να έχουν διεθνείς συμφωνίες κάθε μία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουν να συμμετάσχουν. Εμείς ασχολούμαστε με το θέμα αυτό από τον Ιούλιο του 2017. Υπάρχουν ε, συμφωνίες με την Αργελή, Αλγερία, ε, Ιορδανία και Λίβανο και τελειώνουμε με το Μαρόκο. Τώρα τη συμφωνία. Το Κοινοβούλιο έχει λάβει αυτές τις ε, συμφωνίες ατύπως. Λείπει ακόμα η συμφωνία με το Μαρόκο, όπως σας είπα. Η νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μας είπε να μην πάρουμε ακόμα θέση. Θα περιμένουμε λοιπόν μέχρι να έχουμε και τη συμφωνία του Μαρόκου, αλλά καταρχήν συμφωνούμε απόλυτα να εγκρίνουμε αυτές τις συμφωνίες, ούτως ώστε να γίνει λειτουργικό το πρίμα από την 1η Πρώτου του 2018. Σας ευχαριστώ. Και ο κύριος Ζουρίνι έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε καλές ειδήσει ε, σε ό,τι αφορά την εκτέλεση αυτού του προγράμματος για τη Μεσόγειο. Προβλέπονται πάνω από 400 εκατομμύρια. Και γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να, να παρακολουθήσουμε τι θα γίνει σε ό,τι αφορά τα μέσα αυτά, κατά πόσον θα υπάρχουν, ε, θα επιτευχθούν οι στόχοι τη επιστική ασφάλεια κτλ. Αλλά λόγω τη αλλαγή του κλίματο θα υπάρξουν στρατηγικά προβλήματα, τα οποία θα γίνονται όλο και πιο πιεστικά. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μα ε, ότι ε, δεν θα πρέπει να υπάρχουν πλέον καθυστερήσει και σε ό,τι αφορά τι εργασίε του Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να τονίσουμε τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου που βελτίωσαν σημαντικά το πρόγραμμα σε σχέση με το αρχικό σχέδιο. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω τις συμφωνίες ε, με τρίτες χώρες, ε, Αλγερία, Ιορδανία, Λίβανος, με όσο πιο πολλές ε, χώρες γίνεται. Θα πρέπει το Κοινοβούλιο να μην καθυστερήσει υπέρ διαδικασία αυτή. Αλλά θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερω ότι μπορούμε να βελτιώσουμε σε ό,τι αφορά τι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο καταρχά, τι προτεραιότητε σε ό,τι αφορά την ε, χρηματοδότηση και στη συνέχεια και πρακτική να μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε και στην πράξη ε, την καινοτόμα έρευνα. Αυτά λοιπόν είναι καλά νέα και δεν θα πρέπει να καθυστερήσουμε περαιτέρω τη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρο. Η πλήρη υποστήριξη λοιπόν από όλε τι πλευρέ, από όλου του συναδέλφου. Και τώρα θα ήθελα να ζητήσω του εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την κυρία Κριστίνα Ρούσο, διευθύντρια στην ε, Γενική Διεύθυνση Έρευνα, θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλου. Χαίρομαι ιδιαίτερω που βρίσκομαι εδώ στην Επιτροπή 3 σήμερα το πρωί για να σας αναφέρω τι γίνεται με τις συμφωνίες πρίμα, τις οποίες, ε, τον, για την οποία την διαπραγμάτευση είμαι υπεύθυνη. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω και εσάς, ε, κύριε Πρόεδρε, την Επιτροπή και την κυρία Σακοράφα για την σπουδαία δουλειά που έγινε. Σπουδαία δουλειά για την έγκριση της βασικής πράξης για το πρίμα και χαίρομαι ιδιαίτερος που η συγγήτρια διορίστηκε η κυρία Σακοράφα για τις συμφωνίες αυτές. Νομίζω ότι όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου εξέφρασαν τη σημασία της ε, συμφωνίας, των συμφωνιών πρίμα και σε ό,τι αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη και την καινοτομία, σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των ε, αιτίων της μετανάστευσης, δημιουργίας θέσης εργασιών και ε, πρόθεση της διπλωματίας επιστημονικής ε. Ε, διπλωματία. Αναγνωρίζουμε τη σημασία των συμφωνίων αυτών. Όπω ξέρετε, βασική πράξη του πρίμα εγκρίθηκε πέρσι τον Ιούλιο στην παρούσα, μάλλον στην φάση τη ε, έγκριση τη βασική πράξη, ξεκινήσαμε και τι επίσημε διαπραγματεύσει για τι συμφωνίε πρίμα. Χαίρομαι ιδιαίτερως που σας αναφέρω ότι αυτέ. Ε, οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν με επιτυχία με τέσσερις από τις χώρες τις οποίες χρειαζόμαστε για διεθνή συνεργασία. Με την Ιορδανία, 10 Ιουλίου ξεκίνησε η συμφωνία με την Ιορδανία και η υπογραφή προβλέπεται στο Παγκόσμιο Φόρουμ Επιστήμης τον Νοέμβριο, 10 Νοεμβρίου. Και επισημαίνω και αυτά που είπε και ο κύριος Ρούμπιχ για τη σημασία του φόρουμ αυτού και το γεγονός ότι μπορούν ε, οι χώρες της Μεσογείου να εμπλακούν πιο πολύ σε θέματα επιστήμης και οι διαπραγματεύσεις με την Αλγερία ολοκληρώθηκαν πολύ γρήγορα τάχιστα 11 Ιουλίου συγκεκριμένα. Ξεκίνησε στο Αλγέρι τότε η διαπραγμάτευση, η συμφωνία ήταν γρήγορε λοιπόν οι διαπραγματεύσει και ολοκληρώθηκαν στι 18 Ιουλίου. Η συμφωνία με τον ε, Λίβανο ξεκίνησε εδώ στι Βρυξέλλε 18 Ιουλίου. Για την Αίγυπτο πήγαν λίγο, κάτσαν λίγο παραπάνω τα πράγματα, αλλά και πάλι ε, ξεκίνησε στις 28 Ιουλίου όπως ε, ανέφερε και η κυρία Γιούσο η νομική υπηρεσία θα πρέπει να εξετάσει ε, τις συμφωνίες ε, αυτές. Δεν υπάρχουν όμως κρυμμένες εκπλήξεις, γιατί οι συμφωνίες περιλαμβάνονται και ακολουθούν τη βάση της βασικής πράξης, του πρίμα. Ελπίζω λοιπόν αυτή η εξετασία από την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου να ολοκληρωθεί γρήγορα και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τάχιστα. Θα επανελθώ στο Μαρόκο στο τέλο τη παρέμβασή μου. Θα ήθελα μόνο να πω ότι βάσει των επιτυχών αυτών των διαπραγματεύσεων με τι τέσσερι αυτέ χώρε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 11 Αυγούστου τις προτάσεις για απόφαση του Συμβουλίου για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή όπου είναι εφαρμοστές αυτές τις συμφωνίες και των συμπερασμάτων ε, το της σύναψης των ε, συμφωνιών με τις χώρες αυτές. 25 Σεπτεμβρίου το Συμβούλιο ενέκρινε την υπογραφή εκ μέρους της Ένωσης των Συμφωνιών Πρίμα και οι συμφωνίες αυτές ε, υποβλήθηκαν τα Χιστάν προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και όπως είπατε κύριε Πρόεδρε, τώρα αυτό που επήγει είναι η συνένεση του Κοινοβουλίου προτού το Συμβούλιο είναι σε θέση να εφαρμόσει τις αποφάσεις αυτές και επίσης όπως αναφέρατε είναι πάρα πολύ σημαντικό η διαδικασία αυτή να γίνει με ταχύς ρυθμούς προκειμένου οι χώρες αυτές να μπορέσουν να συμμετάσχουν στον κόσμο του πρίμα εξ αρχής ως ισότιμοι εταίροι το οποίο αποτελεί και το στόχο της πρωτοβουλίας πρίμα. Πριν κλείσω, να πω δύο λόγια για το Μαρόκο. Οι διαπραγματεύσει με το Μαρόκο έλαβαν χώρα και αυτές. Εγώ μετέβησα στο Ραμπάτ δύο φορές. Ως τώρα. Συμφωνήσαμε επί όλων των όρων της συμφωνίας πρίμα, πέρα από τη ρήτρα εδαφικότητα, το οποίο συνδέεται με ένα ευρύτερο πολιτικό ζήτημα, το οποίο φυσικά έχετε υπόψη σας. Ολοκληρώνουμε λοιπόν τις διαδικασίες και τις συζητήσεις για το συγκεκριμένο αυτό θέμα της εδαφικότητας, της εδαφικής μάλλον εφαρμογής της συμφωνίας και πιστεύω ότι δεδομένη τη γενική συζήτηση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Μαρόκο θα πάρει λίγο παραπάνω η όλη διαδικασία. Όπω σα προτείναμε λοιπόν, θα θέλαμε να προχωρήσουμε με τις τέσσερις αυτές συμφωνίες Ιορδανία, Αλγερία, Λίβανος και ε, Αιγυπτός χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Μπορείτε να υπολογίζετε και σε μένα και σε όλους μου τους συναδέλφους ότι θα συνεχίσουμε να τα δραστηριοποιούμαστε και να είμαστε ενεργοί στη συζήτηση με τον Μαρόκο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ με τον κύριο μου. Ευχαριστώ για την πολύ αισιόδοξη ομιλία της. Η κυρία Σακοράφα έχει το λόγο για να συνοψίσει τη συζήτησή μας και για να εκφράσει παρατηρήσεις. Μου επιτρέψετε καταρχήν κύριε Πρόεδρε να μπορέσω να απαντήσω στον κύριο Μαριά σε κάποιες ενστάσεις και απορίες που έχει εξ αρχής και αυτές έχουν να κάνουν με την ε, μικρή συμμετοχή καταρχήν των χωρών όπως εκείνος διαπίστωσε. Θα ήθελα να του πω ότι μόνο αυτές οι χώρες δεχτήκαν μέχρι στιγμής να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία, ότι δεν συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ΜΚΟ και ότι η Τουρκία είναι συνδεδεμένη με τον ορίζοντα 2020 και δεν γίνεται αλλιώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, με ικανοποίηση θα έλεγα ότι υπάρχει, διαπιστώνω ότι υπάρχει κοινή αντίληψη των πολιτικών ομάδων για την αναγκαιότητα αφενό τη έγκριση των σχετικών διεθνών συμφωνιών επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία και αφετέρου τη επίσπευση σχετική νομοθετική διαδικασία. Θέλω να ολοκληρώσω τη σημερινή μου παρέμβαση με μια δημιουργική προτροπή. Όπω γνωρίζετε, το πρίμα απευθύνεται σε ιδρύματα ανώτατη εκπαίδευση, ερευνητικού φορεί, επιχειρήσει του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως μεγέθους και λοιπούς φορείς που δραστηριοποιούνται στα παραπάνω θέματα και θα περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο την υλοποίηση έργων διεθνούς συνεργασίας. Σας καλώ προσωπικά και ανεξάρτητα από το αν η χώρα σας μετέχει στο πρίμα να συμβάλλετε δυναμικά στην ενημέρωση όλων των δυνητικά δικαιούχων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και των αντίστοιχων φορέων από τις υπόλοιπες χώρες που μετέχουν στο πρίμα. Αποτελεί στοίχημα για όλους μας αυτή η πρωτοβουλία να υπηρετήσει αποτελεσματικά τους σκοπούς για τους οποίους υιοθετήθηκε, ώστε καινοτόμα ερευνητικά έργα να πάρουν σάρκα και οστά και να εξασφαλιστεί για νέα χρηματοδοτική συνέχεια και στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ σας ευχαριστώ. Η προθεσμία για τροπολογίες 20 Οκτωβρίου. Έχουμε μια εβδομάδα πάνω κάτω. στο τέλος της ημέρας, μέχρι τις, α, το κλείσιμο των γραφείων. Αυτά είναι για τις τροπολογίες. Βιαζόμαστε πάρα πολύ σε αυτό το πρόγραμμα. Και τώρα περνάμε από ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα σε ένα πολύ σημαντικό άλλο θέμα. Εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αναδιατύπωση και κοινοί κανόνες της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αναδιατύπωση. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε να κάνουμε το πακέτο καθαρής ενέργειας. Ξεκινήσαμε την τελική συζήτηση πια για τέσσερις νομοθετικές προτάσεις. Έχουμε 2.820 τροπολογίες. Καθώς και τροπολογίες στο σχέδιο έκθεσης του εισηγητή. Βάζουμε όλες τις τροπολογίες μαζί. Είναι 2.820 οι τροπολογίες. Ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση για τα θέματα αυτά. Επίσης έχουμε άλλες δύο προτάσεις, το ACER, Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωση, και ετοιμότητα για την μετώπιση του κινδύνου στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Έχουμε δύο εισηγητές για τα τέσσερα αυτά κείμενα. Ο κύριο Καρίντσι είναι ο πρώτος εισηγητής. Έχετε το λόγο. Καλημέρα πρόεδρε σε όλους. Ως είπε σωστά ο πρόεδρος, για αυτά τα δύο πρώτα νομοθετήματα έχουμε σχεδόν φτάσει στι 3.000 τροπολογίες. Φυσικά οι τροπολογίες αφορούν κυρίως τα ίδια θέματα. Δεν είναι mission impossible λοιπόν, δεν είναι αδύνατη αποστολή το να τις ε, ομαδοποιήσουμε. Οι περισσότερες τροπολογίες πηγαίνουν προς την κατεύθυνση που πρότεινα αρχικά. Δηλαδή είναι να καταστήσουμε λειτουργικές τις αγορές, να περιορίσουμε την παρέμβαση να περιορίσουμε τις ε, στρεβλωτικές επιδοτήσεις και να μειώσουμε τελικά το κόστος της ε, ηλεκτρικής ενέργειας στα, στους καταναλωτές, δηλαδή νοικοκυριά και ε, άτομα. Υπάρχει ένα βασικό θέμα που έχουμε. Θα πρέπει να προωθήσουμε την αγορά, να τη στρέψουμε προς μια συγκεκριμένη τεχνολογία. Μπορώ να μιλήσω και γερμανικά. Για να μην ερμηνεία. Intervention Well, you will start from the very beginning. Ναι, να ξεκινήσετε από την αρχή. Να ξεκινήσω από την αρχή. Μάλιστα. Και τότε θα έχετε και τρία λεπτά. Do we have anything? Nothing. Es funktioniert nicht. Δεν λειτουργεί. Nein, nicht. Is anything working? I'll speak in Latvian. Maybe the Latvian booth. Μήπως να μιλήσω λιδονικά. I'll try once again. I'll continue in English. Is it coming through? Ίσο, με τα αγγλικά και βλέπουμε. Σας ε, μεταφράζουν? Ακούτε τη διερμηνία στα γερμανικά? So what shall we do, Chair? Ε, aber wenn ich auf Deutsch ε, spreche... Ναι, άμα μιλήσω στα γερμανικά θα βγουν στα αγγλικά τα... για τους άλλους. Wenn es auf Deutsch geht, kommt das Englische durch. Εντάξει, θα προσπαθήσω να τα πω στα γερμανικά τότε. Α, αγγλικά. Και αγγλικά. Όλε οι γλώσσε φυσικά δεν τίθενται. Κριστιανέ, τι προτιμά, ε, γερμανικά ή αγγλικά. Αγγλικά, αγγλικά θα μιλήσω, είναι απλούστερο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα, συνάδελφοι. χιλιάδες τροπολογίες έχουμε. Γενικά ε, κινούνται προς τη δική μου κατεύθυνση. Υπάρχει ένα βασικό θέμα που θα πρέπει να απαντήσουμε. Θα πρέπει ο νέος σχεδιασμός της αγοράς να προσανατολιστεί προς μια ε, συγκεκριμένη τεχνολογία. Θα πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερος. Έχουμε πολλές τροπολογίες από συναδέλφους που τονίζουν το ρόλο της αποθήκευσης των προμηθευτών Ηλεκτρική ενέργεια, ανάλογα με τη ζήτηση κτλ. Το βασικό που πρέπει να κάνουμε είναι να λειτουργεί η νομοθεσία στο μέλλον. Γιατί κανένα από εμά ε, δεν θα μπορέσει να προβλέψει σήμερα ποιες τεχνολογίες θα αναπτυχθούν, ποιες θα είναι οι πιο ανταγωνιστικές. Μπορεί, ας πούμε, να έχουμε τρομερές ε, πρόοδους σε κάποιες συγκεκριμένες ε, τεχνολογίες, ας πούμε, ε, τεχνολογίες υδρογόνου κτλ. Δεν έχω ιδέα. Το βασικό θα είναι να κάνουμε το παν, ούτω ώστε όλες οι τεχνολογίες, οι καλύτερες, να λειτουργούν και να μας δώσουν τελικά μια προσέγγιση τεχνολογικά ουδέτερη. Ο βασικός στόχος είναι, εάν λειτουργούν σωστά οι αγορές, δηλαδή έχουμε, αν έχουμε πραγματικό ανταγωνισμό, οι αγορές με τις νέες τεχνολογίες θα μπορέσουν να λειτουργήσουν και να χρησιμοποιήσουν και τις ε, καλύτερες, ας πούμε, ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εγώ θα έλεγα όμως να μην προωθήσουμε τις ΑΠΕ, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις αγορές να προωθήσουμε και θα ακολουθήσουν οι ΑΠΕ. Να μην στοιχηματίσουμε ήδη από τώρα υπέρ μιας α ή β τεχνολογίας. Εγώ αυτή την άποψη έχω. Υπάρχουν διάφορα θέματα, λίγα όμως, που ε, είναι διασκορπισμένες οι απόψεις μας, τα ROC, τα Περιφερειακά Λειτουργικά Κέντρα. Εγώ προτείνω να τα πούμε Περιφερειακά Συντονιστικά Κέντρα και πολλοί συνάδελφοι συμφώνησαν. Το βασικό όμως ερώτημα είναι, θέλουμε μια πιο ευρωπαϊκή προσέγγιση ή απλώς μια προσέγγιση εθνική ως προς, τους, ως τα συστήματα ε, μεταφοράς της ενέργειας. Ε, το θέμα είναι να μην τρεμοπέζουν τα φώτα, έτσι. Να έχουμε μια σταθερή συχνότητα, 50 με Hz. Υπάρχει ένα βασικό στοιχείο διασυνοριακού εμπορίου όμως. Τι γίνεται όταν ένας ε, ε, μεταφορέας ενέργειας, ας πούμε, συγκρούεται με έναν άλλον ή στο σημείο, ας πούμε, που αλλάζει και περνάμε από τον ένα στον άλλον ε, διαχειριστή συστήματος. Το δεύτερο θέμα που έχουμε είναι τα πρότυπα επιδόσεως για τις εκπομπές το capacity mechanism, το μηχανισμό δυναμικού, το 550 που συζητάνε όλοι. Εδώ έχουμε πάρα πολλές διαγραφές, δηλαδή κανένα όριο. Έχουμε αυτούς που λένε όχι 550 αλλά 450, έχουμε αυτούς που λένε όχι 450 αλλά 350, έχουμε αυτούς που λένε ότι δεν αφορούν, δεν μπορούν να εφαρμοστούν στις ε, στρατηγικές, ε, στα αποθέματα και ορισμένοι, ορισμένοι λένε μόνο για τις εισαγωγές. Εμείς λοιπόν ως ε, Κοινοβούλιο καλύψαμε όλο το πεδίο. Θα πρέπει να συζητήσουμε και να βρούμε μια λογική προσέγγιση. Κάποια κράτη-μέλη συμπαράγουν και επομένως είναι εξαρτώμενα το, άλλο, το ένα από το άλλο. Ε, ορισμένα άλλα εξαρτώνται από την πυρηνική ενέργεια, άλλα έχουν πολλές ΑΠΕ, άλλα χρησιμοποιούν περισσότερο φυσικό αέριο. Επομένως, έχουμε πολλές διαφορετικές απόψεις και θα είναι μεγάλη πρόκληση να βρούμε μια κοινή ε, γραμμή. Και θα δούμε και μετά τι θα γίνει και με το Συμβούλιο στους τριμερείς διαλόγους. Όταν πάτε τώρα στην οδηγία υπάρχει το θέμα των αριθμιζόμενων τιμών Καταλαβαίνω πλήρως και αναγνωρίζω ότι σε διάφορα κράτη-μέλη υπάρχουν διαφορετικές καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές. Σε ορισμένα κράτη της Ευρώπης, σε μέρη της Ευρώπης, ε, δεν υπάρχει καμία ρύθμιση για τα νοικοκυριά και για τις ε, εταιρείε. Ε, υπάρχει απορρίθμιση και ανταγωνισμός πολύ μεγάλος σχετικά χαμηλέ τιμέ για τα νοικοκυριά, ας πούμε, για την ηλεκτρική ενέργεια σε σχέση με άλλα μέρη τη Ευρώπη. Ε, ε, σε μερικέ περιοχέ λειτουργεί αυτό, σε άλλε περιοχέ τη Ευρώπη έχουμε ρυθμιζόμενε τιμέ, καθορισμένε. Η ιδέα είναι να μην τιμωρήσουμε κανένα σύστημα το οποίο έχει φυσικά ρυθμιζόμενε τιμέ, γιατί οι ρυθμιζόμενε τιμέ συχνά είναι αποτέλεσμα έλλειψη ανταγωνισμού, έλλειψη διασύνδεση. Εάν απορριθμίσει, α πούμε, αν δεν έχει το σωστό ανταγωνισμό, τότε μπορεί οι τιμέ να αυξηθούν. Εγώ αν είμαι μονοπόλιο ας πούμε και με απορριθμίσεις, ε, φυσικά θα αυξήσω την τιμή μου έτσι, και μόνο ο ανταγωνισμός θα την κρατήσει κάτω. Αυτό που σημαίνει, που είναι σημαντικό είναι να κρατήσουμε την ε, πορεία, δηλαδή θα πρέπει να πάμε προς την απορρίθμιση των τιμών, αλλά χωρίς να τιμωρήσουμε ας πούμε, τμήματα της αγοράς. Για να απορριθμίσεις θα πρέπει να είσαι σίγουρος ότι όλα τα υπόλοιπα στοιχεία υπάρχουν έτσι, στην εξίσωση. Ε, ξεπέρασα τα πέντε λεπτά μου, σχεδόν είμαι στα έξι. Κάναμε την πρώτη συνάντηση σκιωδών, είμαι ανοιχτός, ή θα είναι δύσκολη, αλλά είμαι πεπισμένο ότι στο Κοινοβούλιο θα φτάσουμε σε κοινή προσέγγιση που τελικά θα είναι υπέρ τη ανάπτυξη ανταγωνιστικών αγορών στην ηλεκτρική ενέργεια. Ευχαριστώ. Πολύ. Τονίσατε με πάρα πολύ ακρίβεια όλα τα σημαντικά θέματα στην εισήγησή σας εκ μέρους η κυρία Βέρνερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το είπατε για τους... Έχουμε 3.000 τροπολογίες περίπου επιτάπητος, αλλά είμαι πεπισμένη ότι θα καταρθώσουμε να βρούμε μια καλή θέση για το Κοινοβούλιο τα βασικά ζητήματα, για παράδειγμα, σε τη φέρει περιφερειακά κέντρα, σε ό,τι αφορά την ίδρυση μιας ευρωπαϊκής εντότητας για τους διαχειριστές των δικτύων και σε ό,τι αφορά τους μηχανισμούς ε, ικανοτήτων. Σε όλα αυτά συμφωνώ με τον εισηγητή και τους κοιόδης. Σε ό,τι αφορά το, το κέντρο περιφερειακού συντονισμού θα πρέπει να έχει μια αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων σε λίγους αλλά κέρια σημασίας για την περιφερειακή διάσταση και αυτό που είναι σημαντικό να μην υπάρχει παράλληλη καινούργια δομή σε ό,τι αφορά τον συντονιστή της ε, περιφερειακής ασφάλειας δηλαδή. Κύριε Καρίντς, το τονίσατε και εσείς σε αυτό, θα πρέπει να υπάρχουν επικαλύψεις και σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές, την ευρωπαϊκή εντότητα. Οι τροπολογίες μας κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. και οι μικροί διαχειριστές θα πρέπει να μπορούν να είναι μέλη του DSO. Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες για τις αγορές ικανότητας, παρέχουν και αυστηρούς κανόνες για την εισαγωγή τους. Δυστυχώς πιστεύω ότι κάπως έχει καθυστερήσει και τελματώσει η εξέλιξη σε διάφορα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να υπάρχει σαφή διάκριση μεταξύ των μέτρων ε, των εσωτερικών για την αγορά που στρεβλώνουν την αγορά και τέτοια μέτρων που είναι εκτός της αγοράς ως αποθεματικό. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι πολλά κράτη δεν έχουν αποφασίσει προς τα που θα κινηθούν και τι μηχανισμούς ικανότητας θα εισαγάγουν. Σε ό,τι αφορά το Just Transition τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το σκέλος αυτό σε ό,τι αφορά το μηχανισμό, τους μηχανισμό εκανοπτήτων, η αγορά θα πρέπει να απαλλαγεί από τον άνθρακα, αλλά θα πρέπει να είναι και δίκαιοι όροι για τους εργαζόμενους στις διάφορες περιοχές και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αλλαγή, την τρατική αυτή αλλαγή σε διάφορες περιοχές θα πρέπει να γίνει και με πρόγραμμα και σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα και έχω προβλέψει σχετικό άρθρο η ενεργειακή αυτή καμπή χωρίς την υποστήριξη των καταναλωτών δεν πρόκειται να πετύχει και γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό η προστασία των καταναλωτών να ενισχυθεί ως σημείο στην, ε, στο κείμενο. Ύστερα, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αξισορρόπησης, πιστεύω ότι είναι λάθος να καταργηθεί η, προ, η προτεραιότητα τροφοδότηση στο δίκτυο. Νομίζω ότι οι μικρές ε, εγκαταστάσεις θα πρέπει σίγουρα να λεφθούν υπόψη. Προσβλέπω σε μια καλή συνεργασία και με εσά, κύριε Κάριντς, και με τους άλλους εισηγητές και θα ήθελα να τονίσω ότι για μένα προέχει η ενδελάχεια και όχι τόσο η ταχύτητα. Γιατί μιλάμε για τη μεταρρύθμιση όλου του κλάδου παροχής ενέργειας και τη ρύθμιση των αρχών. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται προφανώς χρόνος για να ολοκληρωθεί σωστά αυτή η εργασία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Από την, το ECR. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ένα γενικό σχόλιο Ήδη είχαμε ε, την πρώτη συνάντηση των εισηγητών, έχω διαβάσει τροπολογίες και βλέπω δύο δυνητικούς κινδύνους. Αυτό ισχύει στη σκέψη μας για το πώς θα έπρεπε να ρυθμίσουμε την αγορά ηλεκτρισμού, ηλεκτρικής ενέργειας στο μέλλον. Πρέπει να αποφύγουμε τα δύο άκρα. Το ένα άκρο θα ήταν η τάση να βρούμε μια ιδανική αγορά η οποία θα αυτορυθμίζεται. Να μην υπάρχουν παρεμβάσεις, εξωτερικές παρεμβάσεις. Ε, μια τέτοια ιδανική αγορά θα είχε ως σκοπό να βρει από μόνη της τις σωστές λύσεις. Στη, στο παρελθόν στην Ανατολική Ευρώπη ο Χάιφον Χάιεκ και άλλοι πίστευαν αυτό. Αλλά τώρα ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν ιδανικές αγορές. Αυτός είναι ένας κίνδυνος τον οποίο πρέπει να αποφύγουμε. Και ο άλλος ε, κίνδυνος ε, είναι μια μια μεσιανιστική προσέγγιση, μια ουτοπία. Δηλαδή να αντιμετωπίσουμε το πακέτο σαν μια τελευταία ευκαιρία να σώσουμε την ανθρωπότητα από μια καταστροφή, από την κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή βεβαίως είναι σημαντική και τα θέματα της αγοράς είναι σημαντικά, αλλά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε ε, ρεαλιστικά. Πρέπει να δούμε ποια είναι η τεχνολογική πρόοδος. Βεβαίω πολλά δεν περιλαμβάνονται στο πακέτο. Θα πρέπει να σκεφτούμε και το κοινωνικό κόστος και το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορές στην Ευρώπη, διαφορές οικονομικές ε, και κοινωνικής ανάπτυξης. Υπάρχουν επίσης διαφορές που έχουν να κάνουν με τις διάφορες αρμοδιότητες ε, των περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων και υπάρχουν και άλλες διαμάχες και υπάρχουν και νέα θέματα επίσης. Το θέμα της διαφορετικής αντιμετώπισης των, της ικανότητας ε, και των στρατηγικών αποθεμάτων. Αυτή είναι το μίσα που θα πρέπει να εξετάσουμε με σοβαρότητα. Θα ήθελα να επισύρω την προσοχή σε μια τροπολογία που εγώ κατέθεσα εξ ονόματος της πολιτικής μας ομάδας. Μιλάω ε, για τις ζώνες τιμολόγησης. Μιλήσαμε από τον Διευθυντή Μπόρχαρντ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μας είπε ότι πάρα πολύ συχνά η Κομισιό δεν έχει στην διάθεσή της ορισμένα εργαλεία σε περιπτώσεις κρίσεων. Ε, οι κυκλικές ροές είναι ένα πρόβλημα σημαντικό που εμφανίστηκε πρόσφατα. Αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι ότι η πολιτική μας ομάδα δεν θέλει να εγκαταλείψει πολλές αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ε, περί αυτού πρόκειται σε αυτή την τροπολογία σε ορισμένες ε, περιπτώσεις βλαβών και διακοπών θα πρέπει να έχει βεβαίως ε, ορισμένες αρμοδιότητες η Κομισιόν για τις ζώνες τιμολόγησης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή που άρχισε να εργάζεται σκληρά για να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα με, του τους συμβιβασμούς. Υποστηρίζουμε την προσέγγιση που βασίζεται στην αγορά. Εγώ δεν κατέθεσα ε, τροπολογίες για τους μηχανισμούς ε, για την παραγωγική ικανότητα διότι η προσέγγιση του εισηγητή είναι εδώ και οι ανησυχίες της αγοράς ληφθήκαν υπόψη. Επίσης, γι' αυτό κατέθεσα τροπολογίες υποστηρίζοντας σε μεγάλο βαθμό την προσέγγιση για το dispatch, για την εξισορρόπηση ε, της ευθύνης για το dispatch και την εξισορρόπηση της ευθύνης θα πρέπει να εξαλείψουμε τις εξαιρέσεις. Βεβαίως ε, περιορίζεται η διαφάνεια της αγοράς ε, και δεν ξέρω αν έχουμε πλήρη προσέγγιση για τους μηχανισμούς εξισορρόπησης θα πρέπει την ευθύνη να το δούμε με τρόπο από την άποψη του κόστους ωφέλειας και θα δούμε επίσης την προσφορά των ΑΠΕ. Ε, το να αποφασίσουμε να κρατήσουμε τις εξαιρέσεις αυτές χωρίς να κάνουμε τίποτα για να αναφερθούμε στις ανησυχίες για την ολοκλήρωση της αγοράς. Δεν έχουμε τίποτα μακροπρόθεσμα για την περιφερειακή συνεργασία ψηφέζω ότι τα ρόξα, τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα, δεν ξέρω πώς θα τα ονομάσουν, πρέπει να έχουν αρμοδιότητες λήψεως αποφάσεων. Θα πρέπει να να μην έχει περιορισμούς αυτή η διαδικασία λήψεως αποφάσεων και να έρχομαι μια ισορροπία γεωγραφική, μια χώρα να μην αποφασίζει για όλους, αλλά μια χώρα να μπορεί να λαμβάνει ε, δεσμευτικές αποφάσεις. Σχετικά με το DSO, ε, τις διαχειριστές συστημάτων διανομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει και ο μετασχηματισμός ο ψηφιακός και έχουμε, έχουμε για, για, την, για την τυποποίηση, για το ΆΣΕΡ, έχουμε καταθέσει τροπολογίες αλλά επίσης την ανάπτυξη των smart meters. Πολλές, πολλά κράτη-μέλη έχουν το έχουν ήδη ε, κάνει αυτό, θα πρέπει να τους δώσουμε ε, χρόνο για να κάνουν μια ανάλυση κόστους ωφέλειας. Ε, περιμένω λοιπόν την συνεργασία που θα έχουμε μεταξύ μας. Ευχαριστώ κυρία μου. Ο συνάδελφος Τούρμες από τους Πράσινους. Και εγώ ε, χαίρομαι για τον τρόπο οργάνωσης ε, των συνεδριάσεων των σκιωδών ε, εισηγητών από τον εισηγητή. Προσπάθησε να γίνουν όλα με τρόπο επαγγελματικό. Πρέπει η αγορά να είναι δίκαιη, διαφανής και πέραν των εθνικών συνόρων. Σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να σταματήσουμε όλες τις τρευλώσεις της αγοράς. Το, ο άνθρακας δεν, ε, ε, επίσης ε, το η πυρηνική ενέργεια δεν πληρώνει για την εξάλληψη, για την ενώ υπάρχουν αυτές οι στρεβλώσεις, βρισκόμαστε σε μια αγορά που δουλεύει με στρεβλούς κανόνες. Γιατί έχουμε, έχουμε υπερπαραγωγική ικανότητα γιατί το UEDS έχει αποτύχει και ο άνθρακας δεν πληρώνει ε, για την ρήπανση. Αυτό πρέπει να αλλάξουμε. Να εξαλείψουμε τις στρεβλώσεις στην αγορά. Και ενώ υπάρχουν αυτές οι στρεβλώσεις θα ήταν άδικο να τιμωρούμε τον ένα πόρο που δεν ρηπαίνει, έναν πόρο που ε, δεν αφήνει αρνητική κληρονομιά, τον τιμωρούμε αυτόν τον πόρο, αυτήν την ενέργεια. Αυτό θα ήταν δίκαιο. Χρειαζόμαστε ε, δίκαιο δικαιοσύνη ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην άλλες χώρες. Να κλείσουμε, επειδή έχουμε εξαγωγές ε, από την σερβικό άνθρακα. Αν θέλουμε ηλεκτρονική, ηλεκτρονική ενέργεια από το Μαυροβούνιο που δεν είναι στο ETS, θέλουμε να έρθει στην Ευρώπη. Χρειάζομαστε επίσης ρύθμιση στις αγορές. Πρέπει η αγορά να είναι διαφανής. Αυτό έχει να κάνει με όλες τις υπηρεσίες και για την εξισερόπιση όλων των αποθεμάτων που πρέπει να είναι όσο πιο κοντά ε, στην αγορά και να λαμβάνουν υπόψη την αγορά. Και το τρίτο είναι το, ε, την οικονομική βελτιστοποίηση στην αγορά ηλεκτρισμού πέραν των συνόρων. Πρέπει να καλύψουμε μεγάλες γεωγραφικές περιοχές, αλλά θα πρέπει επίσης να ρυθμιστούν και νομίζω ότι χρειαζόμαστε περισσότερο από συντονισμό στα, στα κέντρα, στα Ρόξ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Έρνστ από την ΚΟΕ. Καταρχάς και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή Άρα σας παρακαλώ, θα είχε νόημα κάποια θέματα και κάποιες τροπολογίες, κάποιες συμβιβαστικέ, μάλλον, να τις, να, να τις ομαδιοποιήσουμε και να τις συζητάμε μαζί. Και παράδειγμα για τις ικανότητες. Έχουμε τόσους παραγράφους που ουσιαστικά μπαίνουν σε μια κατηγορία. Να τις συζητάμε από κοινού. Θα ήταν πιο εύκολο και το κάνουμε και σε άλλες ε, συνεδριάσεις. Τι είναι το πιο σημαντικό για μας τώρα. Τρία στοιχεία. Φυσικά η ασφάλεια τροφοδότησης. Κατά δεύτερον, η πρόσβαση των ατόμων στην ενέργεια. Να μην απρεθεωρητοποιείται κανείς. Και τρίτον, φυσικά, η κλιματική στόχη. Τι νόημα έχει. τα δύο συμβατικά αυτά θέματα να τα συζητάμε, που είναι από τα πιο σημαντικά της θητείας ολόκληρης, το θέμα του κλίματος είναι παράπλευρο. Αυτό το τρίγωνο λοιπόν θα πρέπει να εξετάσουμε. Μόνο αυτό αποτελεί δικαιοσύνη. Όλα τα υπόλοιπα είναι λόγια κενά. Στρέβλωση της αγοράς. Δεν θα το έλεγα όπως ο κύριος Τουρμής, αλλά άμα έτσι τα λέει, εντάξει, συμφωνώ. Πιστεύω ότι τέτοια στρέβλωση τη αγορά δεν επιτρέπεται. Και δεν το εννοώ διανετικά, το εννοώ επί περιεχομένου. Τώρα, σε ό,τι αφορά του μηχανισμού ικανότητα, το συζητήσαμε. Ναι. Ακολουθούμε την κατεύθυνσή σα, αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε τα μεμονωμένα άρθρα, πώ μπορεί να γίνει η λογική οργάνωση. Κάναμε και κάποιε προτάσει. Το θέμα των προσωρινών είναι last resort, τελευταίο. Τελευταία λύση. Και σε αυτό θα πρέπει να συνδεθούν τα υπόλοιπα στοιχεία. Πολλέ είναι οι προτάσει, όπω σα είπα, και θα χαιρόμουν να τα συζητήσουμε επισταμμένω Στρατηγικά από θέματα, και εγώ χαίρομαι. Ξέρω ότι η γερμανική λύση δεν είναι ενδεχομένω η βέλτιστη, αλλά είναι 100 ε, φορέ καλύτερη. Το λέω ξεκάθαρα, δυστυχώ, από πολλέ άλλε λύσει. Προ την κατεύθυνση λοιπόν αυτή θέλω να κινηθώ. Αρχέ ε, τη αγορά Νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε την απελευθέρωση από τον άνθρακα για τα νοικοκυριά χαμηλή κατανάλωση και καλής αποδοτική χρήση τη ενέργεια. Νομίζω ότι αυτά είναι σημαντικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να λεφθούν υπόψη σε ό,τι αφορά την αγορά αυτή. Επίση, πιστεύουμε ότι όλοι οι συμμετέχοντε στην αγορά, όλοι οι παράγοντε τη αγορά, αν υπεύθυνα συμμετέχουν θα πρέπει να συμμετέχουν και στην αγορά ε, εξισορρόπησης. Θα πρέπει να υπάρξει κάποιος συσκελισμός. Θα πρέπει να το διευκρινίσουμε λοιπόν αυτό. Δεν θέλουμε εγκαταστάσεις να εξαιρούνται από την ευθύνη αυτή και από την αγορά λοιπόν εξισορρόπησης. Τώρα, Φυσικά, ξέρετε ότι μα απασχολεί πάρα πολύ αυτή η προτεραιότητα τροφοδοσία στο δίκτυο. Πρέπει να το συζητήσουμε, γιατί στη Γερμανία πετύχαμε τόσο μεγάλη πρόοδο. Τόσο μεγάλη πρόοδο. Δυστυχώ ε, άλλαξε το τέλο η νομοθεσία, λάθο, λάθο ε, μεγάλο. Μέγα σφάλμα. Και ακούμε ότι η Γερμανία δεν θα πετύχει του ενεργειακού τη στόχου, του περιβαλλοντικούς τη στόχου. Εγώ πιστεύω ότι αυτό έχει να κάνει και με το με την αλλαγή αυτή τη νομοθεσία. Να το συζητήσουμε λεπτό λοιπόν ξεκάθαρα. Γιατί πάντα δίνεται προτίμηση στο, στο πυρηνική ενέργεια και στην ενέργεια από άνθρακα. Έτσι έχουν τα πράγματα. Θέλουμε προτεραιότητα λοιπόν τη τροφοδοσία στο δίκτυο για την οδηγία. Θέλουμε να ορίσουμε την ενέργεια του πολίτη θέλουμε το θέμα της ενεργειακής ένδυας να το συζητήσουμε για τα θέματα των ρυθμισμένων τιμών είναι θέμα εθνικό, προστασία του καταναλωτή και να υπάρχει και ένας ανεξάρτητος διαμεσολαβητής. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να ζητήσω το, από τον κύριο Λεβαντόνσκι να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και Κριστιάντη σου εύχομαι καλή τύχη. Καλή τύχη με τις 3.000 τροπολογίες να αναφερθώ σε αυτό το μαγικό αριθμό, το 550, όπως πρότυπο για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Αν ε, υπάρχει πρότυπο ενεργειακό σε αυτό το επίπεδο, σημαίνει κατάργηση της πλειοψηφίας των εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας σε πολλές χώρες. Και στη δική μου χώρα δεν βοηθάει πάρα πολύ θα καταστούμε πιο εξαρτημένοι από εισαγωγές και η εξάρτηση από τις εισαγωγές δεν μπορεί να αποτελεί στόχο της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Και αυτό αποτελεί, αν θέλετε, τιμωρία για κάποιες χώρες, μεταξύ των οποίων και η δική μου. Σε ό,τι αφορά τις προσπάθειές τους να πετύχουν τους περιβαλλοντικούς ε, στόχους. Clean coal technologies, τεχνολογίες καθαρές από άτρακα. Είναι λοιπόν απογοητευτικό αν υπερβάλλουμε σε ό,τι αφορά κάποιες παράμετρους της, του κανονισμού αυτού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Γιούζο τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Κάριντς σε ό,τι αφορά την εργασία του. Οι βασικές με προτάσεις εστιάζονται στον καθορισμό των τιμών κάθε 15 λεπτά. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε την σταθερότητα και ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη που αποζητούν τη διασυνδεσιμότητα. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη και να κοιτάξουμε τον ανοιχτό χαρακτήρα της αγοράς ω αποτέλεσμα των διασυνδεδεμένων δικτύων, πιστεύω ότι αυτό είναι σημαντικό πολύ σε ό,τι αφορά και του ίσου όρου ανταγωνισμού. Η Επιτροπή έχει αφαιρέσει τον dispatch ως προτεραιότητα, αλλά ενδεχομένως να υπάρξει μείωση στο κόστος αυτό του dispatching. Ε, συμπεριλάβαμε επίσης κάποια στοιχεία σε ό,τι αφορά τις τιμές ε, δικτύου που καλύπτουν βασικά έξοδα και τέλη λειτουργία και συντηρήσει, για παράδειγμα, αν είναι καλή η διαχείριση στο πλαίσιο τη εταιρεία. Είναι σημαντικό λοιπόν οι αρχέ αυτέ να οριστούν ε, σε γενικό, συνολικό επίπεδο και όχι να εξαρτώνται από την κάθε υπηρεσία. Σε ό,τι αφορά το όριο διεξοδίου του άνθρακα, θα συμφωνήσω με τον κύριο Λεβαντόφσκι ότι θα πρέπει να είμαστε ε, ευέλικτη και να το αφήσουμε στην διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών προκειμένου να μπορέσουν να προστατεύσουν με τους μηχανισμούς ικανότητας κάποια κέντρα. Σε ό,τι αφορά την ενιαία αγορά έχουμε την αίσθηση ότι οι νομοθέτες θα πρέπει να έχουν λιγότερες αρμοδιότητες προκειμένου στην τελική ανάλυση την πολιτική, την εθνική, να την καθορίσουν τα κράτη-μέλη. Δεν αμφισβητούμε τα συστήματα, των νομοθετή. Αλλά θεωρώ ότι κάποιες από τις αρμοδιότητες των νομοθετή θα πρέπει να είναι λίγο πιο λεπτομερεί, αν θέλετε, σε ό,τι αφορά την ε, τοπική κοινότητα ενέργεια. Αυτό τον ορισμό πιστεύω πρέπει να τον καθορίσουν τα κράτη-μέλη. Και θα πρέπει να είμαστε σε θέση να αποτρέψουμε μεγάλες διακυμάνσεις στην αγορά σε ό,τι αφορά την τιμή της ενέργειας. Σε ό,τι αφορά τώρα το σκέλος της ε, προμήθειας, της παροχής, θα θέλαμε να ενισχυθούν μία σειρά από μέτρα. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντική η διάσταση της διασύνδεσης. Αν δεν υπάρχει 10% διασύνδεση στην Ισπανία, για παράδειγμα, δεν θα είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Τα πηγαίνουμε αρκετά καλά σε ό,τι αφορά τις ανώσιμες ενέργειες. Ωστόσο, νομίζω ότι χάνουμε μεγάλο δυναμικό από τις ανανεώσιμες, αν δεν είχαμε για συναισθημότητα, γιατί δεν θα χρειαζόταν καλά αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη μελητρία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και συμφωνώ απόλυτα με τη φιλοδοξία την οποία εξέφρασε η κυρία Βέρνερ στις ε, τροπολογίες της και αποτελεί έναν από τους πρωταθλητές τη Ήτρας ό,τι αφορά την ενεργειακή φτώχεια, Υπέβαλα λοιπόν τροπολογίες για να προτεθούν οι πολίτες που είναι ενδεείς ό,τι αφορά την ενέργεια. Αυτή η φτώχεια λοιπόν ποτέ δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Τα σα, καθαρά κτίρια θα πρέπει να καταστούν πρότυπο. Και καλώς ορίζω τα σχόλια της ε, Μαρτίνε και της Κορνίλια σε ό,τι αφορά την ενεργειακή ένδυα και Κορνίλια προσπαθούμε να καταρτήσουμε στον ε, φάκελο διακυβέρνηση με ένα σχετικό ορισμό. Αυτό για να υποστηρίξουμε και την περαιτέρω εξέλιξη των ε, τοπικών ε, κοινότητων ενέργειας. Θα πρέπει οι πολίτες να αποτελέσουν τμήμα ενεργό της ενεργειακής καμπής. Μέχρι το 2050 το ίμιση των ευρωπαϊκών νοικοκυριών θα μπορούσαν να παράγουν με ενέργεια 30% θα μπορούσε να προκύψει από την ε, συμμετοχή σε μια τέτοια τοπική ενεργειακή κοινότητα. Θα πρέπει να θέσουμε σωστό επίπεδο φιλοδοξία, γιατί οι πολίτε θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο, στην καρδιά τη ενεργειακή μετάβαση. Καθαρή τιμή και καθαρή ενέργεια σε σωστέ τιμέ για όλου του πολίτε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Κυρία Νίμπλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και να ευχαριστήσω τον εισηγητή, ο οποίο είχε δύσκολο έργο, αλλά νομίζω ότι τα πήγε πάρα πολύ καλά. Του ευχόμαι καλή τύχη. Τέσσερα θέματα θα ήθελα να δείξω και προφανώ θα ήθελα να προσπιστώ και τι τροπολογίε που κατέθεσα. καταρχά μηχανισμοί ικανοτήτων, το οποίο το ανέφεραν πολλοί συνάδελφοι. Εγώ πιστεύω και πρότεινα να υπάρξει διαγραφή σε ό,τι αφορά τα 550 γραμμάρια, γιατί πολύ απλά πιστεύω ότι σε ό,τι αφορά τους μηχανισμούς ικανοτήτων δεν θα πρέπει εδώ να ασκούμε πολιτική για το κλίμα. Έχουμε τους στόχους για το κλίμα και το, εμπόριο των, ε, το σύστημα εμπορία ρήπων. Είμαστε σε φάση διαπραγμάτευση του συστήματος αυτού. Σε ό,τι αφορά του μηχανισμούς ε, ικανοτήτων δεν μιλάμε όμως για το κλίμα. Μιλάμε για την ασφάλεια τροφοδοσία, Μιλάμε για την ευελεξία στην αγορά. Εδώ χρειαζόμαστε λοιπόν ευέλικτε λύσει προσωρινέ λύσει. Γι' αυτό λοιπόν δεν θέλω να γίνει αυτός ο συνδυασμό στο σημείο αυτό. Και νομίζω από πλευρά οικονομικής δεν βγάζει και νόημα. σε ό,τι αφορά και την τιμή για τον καταναλωτή και την κατάργηση ενδεχομένων εγκαταστάσεων. Δεύτερο θέμα, η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Διαχειριστών Δικτύων. Εδώ πιστεύω ότι είναι θετικό το γεγονός ότι υπάρχει πρόταση σε ό,τι αφορά τους διαχειριστές των δικτύων να υποστηριχθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιστεύω ότι αυτό είναι καλό, αλλά θα συμφωνήσω με τον Πέρνερ στο σημείο αυτό. Πιστεύω ότι αν ε, δεν εξαιρέσουμε τις μικρές επιχειρήσεις, ουσιαστικά, ε, αν εξαιρέσουμε τι μικρές επιχειρήσεις, τη χώρα μου θα εξαιρούσαμε το 85% των επιχειρήσεων. Δεν πιστεύω ότι είναι σωστό, δεν στέκει αυτό. Τρίτο θέμα, Ζώνε ε, παροχής και προσφοράς ε, ηλεκτρικού ρεύματο. Ε, εδώ νομίζω ότι αυτό το θέμα αρμοδιότητα. Δεν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει να αποφασίσει το οτιδήποτε σε ό,τι αφορά τι ζώνε ε, ηλεκτρικού. Και τέλο, τελευταίο θέμα, τα περιφερειακά κέντρα ενέργεια. Εδώ, όπω είπαν οι συνάδελφοι, δεν νομίζω ότι υπάρχει οποιαδήποτε ανάγκη να δημιουργηθούν τέτοια κέντρα και νομίζω ότι και αλληλεπικαλύψει και γραφειοκρατία θα προκαλέσει αυτή η ρύθμιση. Δεν βλέπω το λόγο. Διαγραφή ζήτησα και γι' αυτό. Thank you very much, madam. Uh, Mr. Blanco Lopez. Blanco Lopez. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό, αυτός ο νέος σχεδιασμός της αγοράς είναι απαραίτητος για να υπάρξει μία ρύθμιση, γιατί μέχρι στιγμής δεν δίνει σωστές, ε, σωστά μηνύματα για τις τιμές το νέο νομοθέτημα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους νέους ε, φορείς και να τους ενσωματώνει στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας και να λάβουμε υπόψη μας ε, ένα μελλοντικό ενεργειακό μείγμα που θα κυριαρχείται από τις ΑΠΕ. Θα πρέπει να έχουμε μακροπρόθεσμα ασφάλεια, ούτως ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ε, επενδύσεις για καθαρή ενέργεια. Θα ήθελα να σταθώ σε κάποια συγκεκριμένα σημεία για τους μηχανισμούς δυναμικού. Το ηλεκτρικό μείγμα που θα βασίζεται στις ΑΠΕ δεν θα πρέπει να είναι η δικαιολογία, ούτω ώστε να κάνουμε επενδύσει σε μολυσματικές πηγές ενέργειας. Θα πρέπει να έχουμε αυστηρά μέτρα και μόνο ως τελευταία ε, καταφυγή να χρησιμοποιούμε αυτούς τους μηχανισμούς. Είναι λάθος να ακυρώσουμε την, προτεραιότητα, την αποστολή ενέργειας κατά προτεραιότητα και την χρήση των ΑΠΕΚΙ. Ε, γιατί η πρόταση ενέργεια ε, της Κομισιόν είναι πάρα πολύ συντηρητική. Τουλάχιστον θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες των μικρών εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ΑΠΕ, καθώς και τις εγκαταστάσεις επίδειξης που δεν μπορούν, απλής επίδειξης δηλαδή, ε, που δεν μπορούν να ανταγωνιστούν στην αγορά. Δεν θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω μολυσματικών ε, πηγών ενέργειας ε, εις βάρος των καθαρών πηγών ενέργειας. Πρέπει να αναγνωρίσουμε επίσης ε, τη σημασία των διασυνδέσεων. Είναι βασική προϋπόθεση για να αναπτυχθεί η εσωτερική αγορά ενέργειας 100% και να είναι και διαλειτουργική, ενσωματωμένη. Η οδηγία αυτή επίση μιλάει για την ανάγκη προστασία ε, των πολιτών σε περίπτωση που είναι εκτεθειμένοι. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την προστασία και την πρόσβαση στην ενέργεια των πολιτών, ε, ειδικά των πολιτών που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια. Ευχαριστώ τον εισηγητή για τη δουλειά που ε, έκανε και, τους, και του εύχομαι καλή τύχη σε αυτή την περίοδο των διαπραγματεύσεων που είναι μπροστά του. Ευχαριστώ. Ο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Μπόρχαρτ, Μονίμω είστε εδώ στην Επιτροπή μα σχεδόν πάντα. Ε, ο εκπρόσωπο λοιπόν τη Επιτροπής από την ε, Γενική Διεύθυνση ενέργεια, έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ακούσαμε σήμερα το πρωί ότι υπάρχουν σχεδόν 3.000 τροπολογίε. Ουφ, θα μπορούσαμε να πούμε. Κάτι δεν πάει καλά, έτσι. Και με την πρόταση τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ίσω και με τι εκθέσει των εισηγητών. Αλλά εγώ δεν θα το πω αυτό. Αντίθετα, πιστεύω ότι αυτό είναι πραγματικά καλό ε, σημάδι, το γεγονός ότι έχουμε τόσες πολλές τροπολογίες, γιατί αυτό δείχνει τη σημασία που αυτό το μεταρρυθμιστικό πακέτο έχει για την οικονομία μας και για τις κοινωνίες μας. Και επομένως, η Κομισιόν καλωσορίζει αυτή την έντονη δουλειά που παράγει η Επιτροπή σας και τα μέλη της για το φάκελο αυτό. Επίση, η Κομισιόν καλασορίζει το γεγονό ότι οι περισσότερε από τις προτάσεις επικυρώνουν τη γενική ιδέα της Κομισιόν το, του να δηλαδή συστηματικά ακυρώνει τα αυτούς φραγμούς ε, στην, στην αγορά ε, μέσω μιας προσέγγιση που θα βασίζεται στην αγορά. Ε, Κύριε Κρασνοδιεύσκη, η ιδανική αγορά βρίσκεται στα βιβλία. Σωστό είναι αυτό, όχι στην πραγματική ζωή. Ακριβώς γι' αυτό προσπαθήσαμε να βρούμε τη σωστή ισορροπία για να ανοίξουμε την αγορά. Να υπάρχει περισσότερος ανταγωνισμός στην αγορά και να έχουμε ε, μία ολοκλήρωση των ενεργειακών συστημάτων, μία ενσωμάτωση και μία διαδραστική σχέση των διαφορετικών ενεργειακών συστημάτων. Αλλά από την άλλη έχουμε και κάποια περιθώρια ασφάλειας. Και το πιο σημαντικό στοιχείο του είναι ο μηχανισμός ε, αποζημίωσης του δυναμικού. Ανταμοιβής δηλαδή για το παραγόμενο δυναμικό. Εδώ υπάρχουν λοιπόν τώρα διαφορετικές απόψεις ε, στην Επιτροπή. Ε, τι γίνεται με τους κλιματικούς στόχους. Να σας πω κάτι ξεκάθαρο. Φυσικά οι στόχοι της, ε, της ε, κλιματικής πολιτικής πρέπει να ενσωματωθούν στο σύστημα. Όλα αυτά που κάνουμε και που βάζουμε επιτάπητος γίνονται για να αναγνωρίσουμε ότι το ενεργειακό σύστημα είναι ένας από τους μεγαλύτερους ρηπαντές, ένας από τους μεγαλύτερους εχθρούς για το περιβάλλον. Και για πρώτη φορά κάνουμε λοιπόν την προσπάθεια να ενσωματώσουμε τις ΑΠΕ στην αγορά. και να εξασφαλίσουμε μια ενεργειακή αποδοτικότητα η οποία γίνεται πριν ακόμα φτάσουμε στις ΑΠΕ. Αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι να στηρίξουμε την κλιματική πολιτική. Υπάρχουν και άλλα εργαλεία. Το ETS, το, ο μηχανισμός ε, εμπορίας εκπομπών, καθώς και τα 550 γραμμάρια, ο κανόνας ας πούμε ε, της αντιστάθμισης, αποζημίωσης. Το είπαμε πολλές φορές. Για μας χρειάζεται αυτός ο περιορισμός, γιατί όπως υπόθηκε ήδη δεν μπορούμε να δώσουμε τέτοια υποστήριξη μέσω αυτού του μηχανισμού στις πιο ε, ρηπογόνες εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Και εδώ υποστηρίζω, υποστηρίζω πάρα πολύ αυτά που είπε η κυρία Βέρνερ. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια σε μια κατάσταση 42 περιοχών που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιώντας άνθρακα. Δεν γίνεται. Θα πρέπει να έχουμε ενεργές πολιτικές, ούτω ώστε να βοηθήσουμε αυτές τις ρηπογόνε περιοχές να φύγουν από, την, από αυτό το φαύλο κύκλο και να τους δώσουμε την ευκαιρία να αναπτύξουν λιγότερο ρηπογόνες ε, εγκαταστάσεις ε, ή και καθόλου ρηπογόνες ε, εγκαταστάσεις και μάλιστα αυτό να γίνει με κοινωνικά αποδεκτό τρόπο. Και εδώ θα ήθελα να καλέσω τα μέλη αυτής της Επιτροπής να συμμετάσχουν σε αυτή την πλατφόρμα που θα ξεκινήσει στις 11 Δεκεμβρίου με την υποστήριξη της, του Προέδρου και της Επιτροπής σας. Σε αυτή την πλατφόρμα θα βοηθήσουμε και οικονομικά αλλά και θα αναπτύξουμε κάποιες έννοιες, κάποιες ιδέες. Θα ξεκινήσει αυτή η πλατφόρμα, ας πούμε, αν είσαστε στο Στρασβούργο το Δεκέμβριο, αν είσαστε ελεύθερη ανάμεσα στις 4 ε, με 6 με 6,5 και 7 ε, να έρθετε σε αυτή την εκδήλωση ε, που θα είναι πολύ σημαντική για αυτό το θέμα. Τώρα, να σταθώ σε κάποια από τα πιο συγκεκριμένα θέματα τα οποία τέθηκαν. Τα ROCs καταρχήν. Δεν, ROC δηλαδή. Δεν είναι σημαντική, σημαντικό το ακρονίμιο. Το να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη O, operational, το γράμμα O, ε, το επιχειρησιακό ή λειτουργικό ήταν λάθος. Γιατί εμείς δεν θέλουμε να παρέμβουμε στην καθημερινή δουλειά των διαχειριστών συστημάτων. Ε, χαιρόμαστε λοιπόν την αλλαγή στο ακρονίμιο που προτείνει ο εισηγητής, να τα ονομάζουμε συντονιστικά κέντρα και όχι λειτουργικά κέντρα. Στο Συμβούλιο συζητάνε ε, τα security centers, τα κέντρα ασφάλειας, άλλο ακρονίμιο, τρίτο. Εμείς θέλουμε την, το ακρονίμιο του εισηγητή του εισηγητή. Δηλαδή, ε, Regional Cooperation Center, λέει τώρα ο μιλητής, δηλαδή ε, περιφερειακά κέντρα συνεργασίας. Coordination, συγγνώμη, συντονισμού, κέντρα συντονισμού. Η κυρία Βέρνε, ο κύριος Κέλλες και ο κύριος Τούρμες μας υποστήριξαν. Μου άρεσε αυτό. ούτω ώστε να ληφθούν περιφερειακές αποφάσεις σε περιφερειακό επίπεδο δεν, μπορούν, να είναι εθνικές αποφάσεις. Τώρα, για τις ζώνες προσφοράς. Έχουμε την άποψη της κυρίας Νίμπλερ. Καμία εμπλοκή της Κομισιόν. Καμία παρέμβαση της Κομισιόν. Και ο κύριος Κρασνοντεύσκη είπε ότι η Κομισιόν πρέπει να έχει αρμοδιότητες σε αυτές τις ζώνες προσφοράς στα bidding zones. Ε, και οι δύο έχουν δίκιο, αλλά νομίζω ότι το πάνε στα άκρα. Αυτό που πρέπει να αναγνωρίσουμε είναι ότι οι ζώνες προσφοράς δεν είναι μόνο τεχνικό θέμα, είναι και πολιτικό θέμα. Και άρα πιστεύω ότι ο συμβιβασμός θα πρέπει να είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, εντονότερη συμμετοχή των κρατών μελών πριν λάβει δράση η Κομισιόν και δει, ας πούμε, τι μπορεί να χρειάζεται σε αυτό το επίπεδο. Τώρα, για το λιανεμπόριο. Δύο με τρεις σύντομε παρατηρήσει. Οι ρυθμιζόμενε τιμέ, η ρύθμιση των τιμών. Να σα πω κάτι ξεκάθαρα. Τίποτα δεν είναι πιο επιζήμιο στο λιανεμπόριο από το να παρεμβαίνουμε και να καθορίζουμε τι τιμέ. Οποιαδήποτε εξαίρεση που επιτρέπουμε σε αυτό θα οδηγήσει σε όλο και περισσότερα προβλήματα και σε όλο και μεγαλύτερη υπόσκαψη αυτής της έννοιας της αγοράς. Δηλαδή. Θα πρέπει να κρατήσουμε ψηλά τη φιλοδοξία και να αφήσουμε την πολιτική έξω από την, ε, το θέμα της ρυθμίσης των τιμών. Επίσης, θα πρέπει να επιβάλλουμε τον ανταγωνισμό και στους ήδη υπάρχοντες φορείς. Έτσι. Είναι ο καλύτερος τρόπος, ο καλύτερος μηχανισμός για να κρατήσουμε κάτω τις τιμές. Τώρα για τους TSO, δηλαδή θα πρέπει οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς να δεχτούν το άνοιγμα της αγοράς και εμείς με τις τέσσερις οργανώσεις των ε, TSO, των διαχειριστών αυτών, έχουμε συνεργαστεί. Ε, ανοίγουμε, θα πρέπει να ανοίξει η αγορά σε όλους τους διαχειριστές. Το θέμα είναι πώς θα τα ρυθμίσουμε όλα αυτά, πώς θα τα κατασκευάσουμε. Εδώ θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις και κλείνει το μικρόφωνο του ομιλητή. Κυρία Γκρίφιν, μία λέξη. Καταρχάς σας ευχαριστώ για την υποστήριξη για τις τοπικές κοινότητες ενέργειας. Συμφωνώ με αυτά που είπατε. Έχουμε πρόβλημα με τη διατύπωση. Δεν είναι τόσο ξεκάθαρο. Και γι' αυτό προσπαθούμε να τη βελτιώσουμε τη διατύπωση. Γιατί υπήρξαν ερμηνείες των διατάξεών μας, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε καταχρήσεις αυτής της έννοιας. Και σας ευχαριστώ που θέσατε αυτή την έννοια ε, με την οποία συμφωνούμε και ιδίως στο σωστό της πλαίσιο. Ευχαριστώ κύριε Διευθυντά για τις ε, επαγγελματικές ε, παρατηρήσεις ε, εκ μέρους της Επιτροπής για τις διάφορες απόψεις των πολιτικών ομάδων. Βεβαίως οι επαγγελματίες και οι εμπειρογνώμονες είναι πάντοτε ευπρόσδεκτοι. Και τώρα θα ήθελα να σας υπενθυμίσω... Α, α ο κύριος Κάριντς πρώτα απ' όλα, για να συνοψίσει όλη τη συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όσους έλαβαν τον λόγο, κυρίως τους κοιόδης εισηγητές. Θα μπορώ να κάνω ένα σχόλιο. Είχαμε την πρώτη συνεδρίαση με μία μισή ώρα μιλώντας για το άρθρο 1 και 2 ε, που είναι το θέμα και το πεδίο εφαρμογής και το άρθρο 2 είναι το θέμα των ορισμών. Βεβαίως ε, δεν θα ασχοληθούμε με κάθε άρθρο ξεχωριστά, αλλά με κάθε θέμα. Και βεβαίως θα δούμε τα θέματα που δεν είναι επίμαχα. Βεβαίως θα υπάρξουν επίμαχα, είμαστε πολιτικοί, υπάρχουν επίμαχα σημεία παντού. Θα δούμε το κάθε θέμα, τους μηχανισμούς, το dispatching, ε, την ευθύνη εξισορρόπησης, συσίζα ε, η Κομισιόν στην Κομισιόν αρέσει αυτό το ακρονίμιο. Θα ασχοληθούμε με κάθε θέμα ξεχωριστά. Δεν, δεν είμαστε τόσο μακριά ημένα από τους δε. Όλοι μιλάνε έχοντας ε, μία έννοια, μία, ε, κάτι που μας απασχολεί. Δεν είμαστε τόσο διαφορετικοί στις απόψεις μας βάσει των ε, πολιτικών μας πεπιθήσεων. Πολύ συχνά οι τροπολογίες μας ε, προέρχονται κυρίως από την περιφέρεια από την οποία προερχόμαστε ως πολιτικοί, από την εκλογική μας περιφέρεια. Και ο λόγος βεβαίως είναι ότι αυτές οι ανησυχίες είναι πραγματικές σε ορισμένα μέρη την Ευρώπη. Οι διασυνδέσεις είναι μια, μια πραγματική ε, πρόκληση για να λειτουργήσει η αγορά. Αυτό έχει να κάνει με τις διασυνοριακές ε, ροές, ε, την ικανότητα που χρειάζεται η απορρίθμιση των τιμών. Αυτά όλα είναι μέρος του πακέτου. Αυτά τα μέλη που προέρχονται από περιοχές που παράγουν ε, άνθρακα, πρέπει να καταλάβουμε τις ανησυχίες τους. Στην δική μου περιφέρεια δεν υπάρχει άνθρακας. Ε, δεν ενδιαφέρομαι για το θέμα αυτό εγώ προσωπικά. Αλλά πρόκειται και για ένα κοινωνικό θέμα, διότι εργάζονται πολλοί στον τομέα και πώς, ε, πώς θα γίνει η μετάβαση. Νομίζω ότι κανείς δεν αμφισβητεί την ιδέα ότι πρέπει να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος, μια μετάβαση. Πώς θα γίνει αυτό. Και αυτό επίσης με τις ζώνες προσφοράς, με το ρόλο της Επιτροπής. Βεβαίως πρόκειται για ένα θέμα τεχνικό, ένα θέμα που βασίζεται στην αγορά και όταν μιλώ για τις ε, κέντρα ασφαλείας και τα κέντρα διανομής όταν, ε, των διαχειριστών ε, συστημάτων διανομής ε, νομίζουν ότι πρέπει να βασιζόμαστε στην τιμολόγηση στους αλγόριθμους. Βεβαίως, δεν νομίζω να υπάρξει κανείς, δεν μιλάει κανείς για μια κομβική τιμολόγηση. Για να δώσουμε βεβαίως τέτοιο σήμα στην αγορά διότι αυτό θα αυξήσει την τιμή της ε, ηλεκτρικής ενέργειας ε, σε ορισμένες περιοχές, κυρίως τις βιομηχανικές που παράγουν μεγάλο μέρος του ΑΕΠ. Θα πρέπει να τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη. Θα πρέπει να βρούμε λύσεις που να εργάζονται. Βεβαίως ε, και η Κομισιόν τονίζει την ανάγκη να βάλουμε την αγορά πρώτη αν δώσουμε τα σωστά μηνύματα, αν εργάζεται καλά, λειτουργεί καλά η αγορά, θα μπορέσουμε να υπηρνικήσουμε πάρα πολλές δυσκολίες. Ε, στην Λετωνία, στη χώρα μου, ε, πριν από 10-15 χρόνια, ήμασταν ε, για στην αέριο και στην ηλεκτρική ενέργεια. Χάρη στα PCIs έχουμε μεγάλες ε, διασυνδέσεις με τους βόρειους ε, γείτονές μας. Έχουμε ένα Northern Pool για μια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και έχουμε ένα ένα spot market και βλέπουμε πώς λειτουργεί και λειτουργεί πάρα πολύ καλά διότι οι όροι είναι πολύ καλοί, οι διασυνδέσεις είναι καλές, οι διάφορες πηγές παραγωγής υπάρχουν σε ολόκληρο το σύστημα και δεν υπάρχουν περιορισμοί στην αγορά, πολιτιστικοί περιορισμοί, φυσικοί περιορισμοί. Είναι, είναι μια ελεύθερη αγορά. Ε, βεβαίως ε, όταν βεβαίως υπάρχει σταθερότητα, οι αγορές πάντοτε διορθώνουν την κατάσταση. Όταν το έχετε αυτό λειτουργεί καλά. Το επιχείρημα είναι ότι μπορεί να λειτουργήσει και θα πρέπει να υπερνικήσουμε ε, τους φραγμούς, τους φυσικούς, τους ε, πολιτικούς, την αντίσταση σε αυτήν την λειτουργία και να γίνουν τα πράγματα καλώς. Είναι κάτι το θετικό και ενδιαφέρομαι πάρα πολύ για όλη αυτή την εργασία που γίνεται με τους... Ε, ε, Ευχαριστώ. Δεν συμμετείχα στη συζήτηση, αλλά εγώ σας λέω ως ακροατής ότι ήταν θαυμάσια συζήτηση. Θαυμάσια για ένα τόσο σημαντικό θέμα. νομίζω από τα πιο σημαντικά για το τέλος της θητείας της ε, Επιτροπής μας. Ευχαριστώ για την ευκαιρία προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στις 11 Δεκεμβρίου του 2017 θα ψηφίσουμε στην Ήτρε. Είναι Δευτέρα. Στρασβούργου, αν θυμάμαι κατά. Ε, να είστε έτοιμοι. Το επόμενο σημείο Α, ήρθατε και στην ώρα σας, κυρία Νίμπλερ. Ευχαριστώ. Πρέπει να ψηφίσουμε στο Στρασβούργο. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Πρέπει να ψηφίσουμε ντε και καλά εκεί. Δεν θα ήταν καλή ιδέα. Γιατί στο Στρασβούργο είμαστε όλοι τόσο απασχολημένοι και θα είναι και η τελευταία ολομέλεια της χρονιάς. Καλύτερα να βρούμε μια άλλη ημερομηνία, όχι στο Στρασβούργο στις Βρυξέλλες καλύτερα. Αυτό σας ε, καλό να κάνετε. Έχει μπει στην ατζέντα μας ε, για το Στρασβούργο, δηλαδή η ψηφοφορία γίνει το Στρασβούργο, εδώ και έξι εβδομάδες. Από αρχή Σεπτεμβρίου το συμφωνήσαμε. Δεν μπορούσαμε να βρούμε άλλη λύση, γι' αυτό το προτείναμε αυτό. Εάν θέλουμε να τελειώσουμε μέσα στο 17, πρέπει να το κάνουμε στο Στρασβούργο. Εάν δεν ψηφίσουμε στο Στρασβούργο, τότε θα τελειώσουμε αναγκαστικά στον, τον Ιανουάριο. Αλλά δεν το θέλουμε. Αρχικά είχαμε πει να έχουμε ολοκληρώσει τέλος Νοεμβρίου, αλλά ήταν αδύνατον αυτό. Γιατί έχουμε ατελείωτες τροπολογίες, πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε. Προσθέσαμε λοιπόν δύο εβδομάδες. Δηλαδή πήγαμε από τέλος Νοεμβρίου, 11 Δεκεμβρίου. Είναι δύο σημαντικές εβδομάδες όπου θα εργαστούμε επί των συμβαστικών τροπολογιών ε, πάνω σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Έχουμε και άλλους φακέλους που θα τους ψηφίσουμε στις 11 Δεκεμβρίου μαζί. Τέσσερα θέματα είναι αυτά που θα ψηφίσουμε στις 11 του μηνός. Καταλαβαίνω το πρόβλημά σας, σωστό είναι αυτό που λέτε. Θέλαμε και εμείς να το αποφύγουμε, αλλά δεν γινόταν. Αν θέλουμε να τελειώσουμε στο 17, είναι απαραίτητο να το κάνουμε στο Στρασβούργο του Δεκεμβρίου. Και τώρα πάμε στο 16. Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναδιατύπωση. Ο εισηγητή μας, Μόρτεν Χέλβεκ Πέρτερσεν. Πρέπει να πω ότι και αυτό το θέμα είναι τμήμα του πακέτου καθαρής ενέργειας και συνδέεται εκ του σύνεγγυς με τους άλλους φακέλους, κυρίως με αυτό που μόλις συζητήσαμε. Η αναθεώρηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και όλα τα θέματα του Άσερ είναι ελενδετα Θέλουμε να επικαιροποιήσουμε τον κανονισμό ασερ Acer για να αντικατοπτρίζουμε τις, τα νέα καθήκοντα που παίρνει ο οργανισμός από που παίρνει, εν περιπτώσει, και να επιτρέψουμε να αλλάξουν οι κανόνες. Έχουμε 412 τροπολογίες. Τυχερός είστε, Μόρτεν. Πολύ λιγότερες ε, τροπολογίες, γιατί ο Κρίστιαν έχει πολύ περισσότερες. Διάφορα θέματα αφορούν οι τροπολογίες και τους, ε, τα καθήκοντα και τους στόχους της, ε, του οργανισμού, καθώς τον τρόπο λήψης των αποφάσεων, την εσωτερική οργάνωση κτλ. Έχετε τον λόγο. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και όντω ε, δίκιο έχετε. Δεν έχουμε τέτοιο συντριπτικό, συνθλιφτικό ρυθμό προπολογιών όπως ο κύριος Κάρινς, αλλά καταρχάς να ευχαριστήσω τους σκιώτες για τη συμβολή τους. Και γενικά να πω ότι είμαι αισιόδοξο. Πιστεύω ότι θα είναι καλό ο κανονισμό. Ήταν πολλέ και επικοδομητικέ ιδέε που ακούσαμε από όλου του κοιόδη. Οι πρώτε δε συναντήσει με του κοιόδη ε, σίγουρα προμηνύουν ε, ζωηρέ συζητήσει, αλλά είμαι βέβαιο ότι θα τα καταφέρουμε. Επισκέφτηκα λοιπόν το Acer πριν από κάποιε εβδομάδε. Μεγάλη μου χαρά. Και τα στοιχεία, τα στατιστικά και τα αριθμητικά καταδεικνύουν ότι όποτε η ενέργεια φτάνει στα σύνορα, ουσιαστικά σταματάει η ροή. Δεν υπάρχει ουσιαστικά ενιαία αγορά στην ενέργεια. Φαίνεται αυτό σαφέστατα από τα στοιχεία. Ότι έχουμε τόσα εμπόδια στα σύνορα και αυτό σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να το καταπολεμήσουμε, να το αλλάξουμε. Αυτό φαίνεται και από την προηγούμενη έκθεση και σε ό,τι αφορά και τις ε, αρμοδιότητες ε, που υπάρχουν. Θα τεθούν πολλά ζητήματα σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες των διευθυντών, ε, σε ό,τι αφορά το άσερ, τα δικαιώματα ψήφου, τη σύνθεση κτλ. Αλλά με βέβαια ότι θα καταλήξουμε σε συμβιβασμού. Θα γίνουν και συζητήσει για περιφερειακά ζητήματα. Και θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι δυνατότητα έχει να λαμβάνει μόνιμες ε, ε, αποφάσεις. Σίγουρα θα γίνει λοιπόν η συζήτηση αυτή και για το φάκελο αυτό και είναι σημαντικό να συντονιστούμε και με το θέμα σχεδιασμού της αγοράς και να υπάρχει και μια συνεκτικότητα, να υπάρχει συνέχεια. Θα γίνουν συγκεκριμένε λοιπόν συζητήσει για το θέμα αυτό. Άρα, Πρόεδρε, εγώ είμαι βέβαιος και αισιόδοξο ότι οι συζητήσεις θα είναι καλές. Να ευχαριστήσω τους κοιόδες για την επικοδομητική στάση που έχουν δείξει τώρα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ αλλά και Πρόεδρο σου. Η κυρία Νίμπλερ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ σήμερα εκπρόσωπω τον κύριο Βέρνερ Λάγκερ, τον συνάδελφο, ο οποίος ε, έχει ε, άλλες υποχρεώσεις σε άλλη επιτροπή και ζητά συγγνώμη που δεν μπορεί να συμμετάσχει. Αλλά μου έχει δώσει σαφέστατες οδηγίε. Καταρχάς, ευχαριστεί τον εισηγητή για τους ε, συναντήσεις των σκιωδών. Η συνάντηση των σκιωδών έλαβε χώρα ήδη την τρέχουσα εβδομάδα και θεωρεί ότι η πρώτη συζήτηση δυστυχώς δεν ε, έχει θέσει το πλαίσιο για σωστές και επικοδομητικές συμβαστικές λύσεις. Και, Κάποια ζητήματα δεν έχουν ακόμα αναφερθεί, δυστυχώς, αλλά εκφράζουμε την απόλυτη εμπιστοσύνη που έχει προς τον εισηγητή και ότι στο Στρασβούργο στην επόμενη συνεδρίαση θα υπάρξει συνταλλαγή απόψε για τα σημαντικότερα στοιχεία της νομοθεσίας. Ο συνάδελφος Λάγκε θέλει να εκφράσει τα βασικά θέματα που απασχολούν το ΕΛΚ επ' ευκαιρία και θα ήθελα να σα παρουσιάσω ποια είναι αυτά τα τέσσερα θέματα. Καταρχά, σε ό,τι αφορά την ευάθυνση τη ενιαία αγορά, θα πρέπει να ενισχυθεί ο Acer. Ωστόσο, η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων θα πρέπει αποκλειστικά να ε, έχει να κάνει με διασυνοριακά ζητήματα ή αμφιλεγόμενες περιπτώσεις. Κατά δεύτερον, το, α, οι αποφάσεις στο Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνονται κατά δύο τρίτα, με δύο τρίτα. Κατά τρίτον, οι αρμοδιότητες μεταξύ Διοικητικού Συμβουλίου, α, Ρυθμιστικού Συμβουλίου και των υπόλοιπων σωμάτων θα πρέπει να διελευκαθούν. Τελευταίο θέμα. Ο κύριος Λάγκεν πιστεύει ότι υπάρχουν οικονομικέ δυσκολίες ό,τι αφορά το Acer, το διαπιστώνει αυτό, αλλά δεν πιστεύει ότι αυτό μπορεί να επιληθεί με επιβολή τελών από τον Acer. Μόνο σε κατεξαίρεση περιπτώσεις θα πρέπει να επιβάλλονται τέλη. Αυτά λοιπόν είναι τα πιο βασικά θέματα τα οποία ο εισηγητής μας, Βέρνερ ο, ο, ο Βέρνερ ε, Λάγκερ, ήθελε να θέσει στα πλαίσια της συζήτησης αυτής, αλλά σίγουρα θα τα προβάλλει και στην επόμενη συνεδρίαση των σκιωδών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει και πρόεδρος. Σαφέστατα τα σχόλια και παρατηρήσεις. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στον επόμενο συνάδελφο, εξ ονόματος των σοσιαλιστών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Και μπορούμε να διαιρέσουμε, αν θέλετε, να κατεργοποιήσουμε τη συζήτηση σε δύο επίπεδα. Αύξηση των αρμοδιοτήτων για τα οποία χρειάζονται αποφάσεις περιφερειακής συνεργασίας και στη συνέχεια τα μεμονωμένα σώματα, διευθυντές, συμβούλιο και το καθεξής. Εγώ υποστηρίζω την αύξηση των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών του οργανισμού. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης όταν ε, υπάρχει θέμα διορισμού περιφερειακών κέντρων και το καθεξής ή άλλου θέματος που έχει να κάνει με την διασυνοριακή διάσταση και είναι κατά παραβίαση των κοινωτικών διατάξεων. Επίσης, ο οργανισμός θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει πληροφορίες από τους παράγοντες της αγοράς για να εκπληρώσει τα καθήκοντά του. Θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να εφαρμόζει τις αποφάσεις του. Υποστηρίζω επίσης την αύξηση και την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας στο σύνολό της. Αυτό μόνο σε καλύτερη λειτουργία της αγοράς μπορεί να οδηγήσει και σε μείωση του κόστους. Τα περιφερειακά κέντρα τα οποία ορίζονται στον κανονισμό αποτελούν έναν τρόπο να το πετύχουμε αυτό. Η αγορά αν είναι όλο και πιο διασυνδεδεμένη και αυτό αποτελεί ένα βασικό όρο για τη λειτουργία τη αγορά. Αλλά υπάρχουν τρία ζητήματα. Ε, έχουμε ακόμα έλλειψη σε ανθρώπινου και οικονομικού πόρου. Πριν από λίγε εβδομάδε. πήγαμε σε Λιμπιουάνα, σε ένα κέντρο εκεί του Acer. σαφώ, λοιπόν υπάρχει έλλειψη πόρων και θα πρέπει η υπηρεσία να έχει επαρκές και προσωπικό αλλά και επαρκή μέσα, υπάρχει κονδύλια για να εκτελεί τα καθήκοντά τη. Άρα λοιπόν θα υποστήριζα ανεχόμενη επιβολή τελών στα πλαίσια της λειτουργίας της αγοράς. Κατά δεύτερον, θέματα ανεξαρτησίας της, ε, του οργανισμού. Και αυτό είναι πολύ βασικό, η ανεξαρτησία για τη λειτουργία του οργανισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του δεν ε, θα πρέπει να υπόκειται καμία πολιτική πίεση και να μην δέχονται πολιτικέ οδηγίε. Επίση, ο διευθυντή θα πρέπει να είναι απόλυτα ανεξάρτητο και νομίζω ότι ο διορισμό του διευθυντή θα πρέπει να αποτελεί αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μία από τι αρμοδιότητε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπω γίνεται και σε άλλου οργανισμού, για να υπάρχει μια σωστή εξισορρόπηση των δυνάμεων. Αν του δώσουμε πιο πολλέ αρμοδιότητε, να έχουν και πιο πολλέ ευθύνε. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να οριστούν αυτά με τον σωστό τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Από το ECR, ο κύριος Χέγκελ, ο αντιπρόεδρος μας. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι πολύ σημαντικό θέμα και αποτελεί μέρος όλου του πακέτου του ενεργειακού ε, στην Ευρώπη είμαστε υπερήφανοι για την ε, κοινή μας αγορά ε, και θέλουμε να προχωρήσουμε περισσότερο στην ενεργειακή αγορά. Βεβαίως, χαιρόμαστε για την περιφερειακή συνεργασία, αλλά μόνο η Σουηδία και η Νορβηγία συνεργάζονται καλά, διότι αισθάνονται την ανάγκη να το πράττουν, παρά τους στόχους διασύνδεση τα κράτη-μέλη ε, διασυνδέονται λίγο, συνεργάζονται λίγο και εργαζόμενοι για το θέμα αυτό. Είδατε ανεξάρτητα του αν ε, μιλούμε για ε, το, τις διάφορες πρωτεύουσες, η μεγάλη πλειονότητα κυρίως οι προστατευτιστές θέλουν λιγότερα. Σας καλώ να αφήσετε κατά μέρος τον προστατευτισμό. Χρειαζόμαστε με έναν οργανισμό πιο ισχυρό για να δημιουργήσουμε μια κοινή ενεργειακή αγορά. Χρειαζόμαστε ε, τα κέντρα, ε, τα περιφερειακά, τα συντονιστικά και επιχειρησιακά για να εργαστούν για την παραγωγή, την διανομή. Μιλάμε για το υψηλό κόστος ενέργειας ε, στην Ευρώπη και βεβαίως θέλουμε πιο ε, καθαρή ενέργεια, πιο φθηνή ενέργεια. Δεν πρέπει να κλείνουμε τους στα σύνορα για λόγους προστατευτισμού. Ε, αλλιώ δεν θα έχουμε ποτέ ανταγωνιστικότητα και ανταγωνιστικές και χαμηλές τιμές για τους καταναλωτές. Ας προοδεύσουμε όλοι προς τον κοινό στόχο να έχουμε μια ενεργειακή ένωση με ένα καλό μείγμα ενεργειακό που ε, θα εξασφαλίζει την ασφάλεια εφοδιασμού καλύτερη, συνεργασία περιφερειακή και ανταγωνιστικότητα με χαμηλές τιμές για όλους τους Ευρωπαίους πελάτες η πρόταση της Κομισιόν παρά μερικά να νομίζω είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ας μην τη στραγγαλίσουμε, ας μην την απορρίψουμε. Και βεβαίως ευχαριστούμε τον εισηγητή, τους κοιόδης εισηγητές και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους συναδέλφους για τη συνεργασία τους, αλλά και να προσθέσω ότι νομίζω ότι δεν μπορέσαμε να συμπληρώσουμε το φάκελο αυτό χωρίς την υποστήριξη του προσωπικού μας και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω το προσωπικό μας για την συνεργασία. Ευχαριστώ. Εκ μέρους των Πρασίνων, ο κύριος Δάβολ Σκρέτς. Καλή η, η, η προφορά. Η προφορά καλή. Καλά. Βρέθηκε κάποιος που ξέρει να προφέρει το όνομά μου. Δεν θα σας απασχολήσω πολύ, συναδελφοί. Ευχαριστώ τον εισηγητή μας για την προσπάθειά του να λάβει υπόψη και τις δικές μου τροπολογίες, όπως αναφέρθηκε και από τους προηγούμενους ομιλητές. Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να αναγνωρίσουμε το δυναμικό και το βασικό ρόλο της νέας πρωτοβουλίας αυτής. Οι πράσινοι ε, είναι συστηματικά υπέρ της ιδέας του οργανισμού. Με τις τροπολογίες μου θα θέσουμε το κατάλληλο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργεί ο Acer. Ε, με τις τροπολογίες λαμβάνουμε υπόψη μας διάφορα στοιχεία, αλλά εδώ θέλω να σταθώ σε ένα ειδικά, πιο σημαντικό. Την πολιτική ανεξαρτησία της, α, του Acer. Να μην εξαρτάται από κανένα δημόσιο ιδιωτικό φορέα. Υπάρχει μια, ένα ιδιωτικό λόμπι που είναι καταχωρημένο στις Βρυξέλλες και λέγεται ε, το Συμβούλιο των ε, Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών. Και υπάρχει μια μακρά πρακτική της παρουσίας αυτού του λόμπι στην, ε, στα όργανα, τα διοικητικά όργανα του Άσερ. Επίσης η παρουσία αυτού του Συμβουλίου και ο πρόεδρος του Άσερ ε, που εκπροσωπεί τις εθνικές, το Σύνοδο των Εθνικών Αρχών είναι το ίδιο άτομο. από το Σεπτέμβριο είναι ένα καινούριο άτομο πάντα ο ίδιος, ε, ο οποίος έχει και, τα δύο, και τις δύο θέσεις, ας πούμε, και τα δύο αξιώματα. Αυτό είναι λάθος. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε τη δυνατότητα να σταματήσει αυτή η πρακτική εξωτερικής επιρροής στον Acer. Έχω υποβάλει διάφορε τροπολογίε προ αυτήν την κατεύθυνση και ελπίζω ότι οι συνάδελφοί μου από τι άλλε ομάδε θα με υποστηρίξουν προ αυτό, προ αυτήν την κατεύθυνση. Το δεύτερο που θέλω να θέσω είναι ότι έχω υποβάλει μια τροπολογία που ζητάω ο διευθυντή τη υπηρεσία του οργανισμού να επιβεβαιώνεται στη θέση του αυτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα κριτήρια, ε, καταρχά, θα πρέπει να έρχεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να απαντάει σε ερωτήσει. Καθώ αυξάνονται οι αρμοδιότητε του οργανισμού, ε, θα πρέπει ε, να ελέγχεται όλο και περισσότερο ε, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ο κ. Σιλικιώτης, παρακαλώ. Ο σκιώδης εισηγητής τη ΓΚΟΕ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Merci. για τη δουλειά που έχει κάνει, καθώς και για τη συνεργασία που είχαμε στην πρώτη συνάντηση των σχεδόν εισηγητών, η οποία κρίνω αυτή τη συνάντηση ήταν αρκετά επικοδομητική, παρόλο που ως ομάδα ε, έχουμε σημαντικές διαφορές με τις θέσεις του εισηγητή. Κατά την άποψή μας, καθώς ο ΕΣΕΡ δεν είναι ευρωπαϊκός οργανισμός, αλλά μια πλατφόρμα συνεργασία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών δεν πρέπει να του δοθούν οι ευξημένε αρμοδίδε που προτείνονται. Για μας είναι ξεκάθαρα πως ο ΕΣΕ δεν πρέπει να διαμορφώνει στρατηγική. Οι ιδιαιτερότητες των κρατών μελών, τα ιδιαίτερα προβλήματα και οι ανάγκε που έχουν είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη. Ιδιαίτερα ενώ η Ένωση αποτυχάνει να αντιμετωπίσει ε, τα σοβαρά προβλήματα ενεργειακού εφοδιασμού που υπάρχουν σε μερικέ χώρε, και ούτε έχει, άρει, έχει συμβάλει ώστε να έρθει η ενεργειακή απομόνωση στην οποία βρίσκονται κράτη και περιοχές της Ένωσης. Εν τούτης, ε, δυστυχώς, οι προτάσεις που αναπτύσσονται στον κανονισμό για αυξημένες αρμοδιότητες των ΕΣΕΡ καταστρατηγούν τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών στη διαμόρφωση της ενεργειακής πολιτικής και υπονομεύουν, ε, κατά την άποψή μας, το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν μέχρι σήμερα οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Ιδιαίτερα προβληματική κατά τη γνώμη μα είναι η πρόταση του άρθρου 43 πω το Διοικητικό Συμβούλιο του Acer θα εγκρίνει στρατηγική για τι σχέσει με τρίτε χώρε. Ο Acer δεν είναι πολιτικό όργανο και δεν πρέπει να λάβει τέτοιε υπερεξουσίε. Η όρη συνεργασία με τρίτε χώρε είναι απόφαση των κρατών μελών και αφορά μονάχα στι σχέσει με εκείνε τι τρίτε χώρε που έχουν υιοθετήσει και εφαρμόζουν το κεκτημένο της Ένωσης στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος κατόπιν σύναψης συμφωνιών με την Ένωση. Δεν μπορεί λοιπόν ο ΕΣΕΡ να αποφασίζει αυθαίρετα βάσει άλλων κριτηρίων για τόσο σημαντικά θέματα. Ολοκληρώνοντα, θα ήθελα να αναφερθώ στο Ρυθμιστικό Συμβούλιο, που είναι και το κύριο όργανο λήψη αποφάσεων του ΕΣΕΡ. Η αντικειμενική λειτουργία του και η αντιπροσωπευτική συμμετοχή όλων των μελών του είναι ζωτική σημασία. Για τον λόγο αυτό, η τροποποίηση προτείνεται στο άρθρο 23 όσον αφορά του κανόνε ψηφοφορία. Για παράδειγμα, πριν χρειαζόταν δύο τρίτα για να περάσει μια απόφαση, τότε τώρα απαιτείται απλή πλειοψηφία. Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη και κατά την άποψή μα υπονομεύει τη λεπτή ισορροπία τη αντιπροσωπευτική συμμετοχή που υπάρχει στον Acer και που πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει, δηλαδή να υπάρχει ισχυρή πλειοψηφία στην ε, διαμόρφωση των αποφάσεων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Διευθυντής Κλάους Τίτερ Μπορχαρτ, έχετε το λόγο κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ και ελπίζω ότι αυτή τη φορά ε, θα είμαι πολύ πιο σύντομος από την πρώτη παρέμβασή μου. Από ό,τι κατάλαβα από τη συζήτηση τη σημερινή ε, και από την ε, καλή εισήγηση είναι ότι πιστεύουμε όλοι ότι μια πραγματική ενεργειακή ένωση θα είναι κάτι όπου θα μπορούμε να αποφασίσουμε για ρυθμιστικά θέματα και για διασυνοριακές καταστάσεις. Εδώ πρέπει να πω ότι ήδη και τώρα ο ρόλος των ρυθμιστών ε, των εθνικών και η συνεργασία με τον Άσερ είναι αρκετά στενή. Και αυτό δεν το αλλάξαμε. Ο οργανισμός, ο Άσερ, ε, θα μείνει βάση της ε, πρότασή μας ε, εκεί όπου θα πρέπει οι ρυθμιστές να βρουν μια συμφωνία με την βοήθεια του Άσερ. Αυτό θα πρέπει να το συμφωνήσουμε όλοι μας εδώ. Τώρα, ο ίδιος ο εισηγητής ανέφερε ένα θέμα το οποίο λείπει από την πρότασή μας. Έκανε τη σύνδεση με τα περιφερειακά κέντρα συνεργασίας και είναι αλήθεια ότι στη δική μας την πρόταση αυτά τα κέντρα ε, δεν αντανακλώνται ε, σε επίπεδο ρυθμιστικό. Και νομίζω ότι θα είναι χρήσιμο να σκεφτεί κανείς με αυτόν τον τρόπο και να προσθεθεί αυτό το στοιχείο που λείπει. Για τα υπόλοιπα, νομίζω ότι η κυρία Μίντλερ, εκ του κυρίου Λάγκε, συνόψισε πάρα πολύ καλά τα βασικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσει αυτή η Επιτροπή. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, διότι θα αφήσω την εργασία σε εσά και ξέρετε πολύ καλά την πρόταση της Κομισιό. Θα ήθελα να αναφέρω δύο πράγματα. Ο κύριος Χόχ, ο οποίος ανέφερε κάτι το σημαντικό, ε, την ε, συλλογή πληροφοριών που χρειάζεται ο Άσερ για την παρακολούθηση της αγοράς και εδώ η κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να ενισχύσουμε ε, την συλλογή πληροφοριών και τις αρμοδιότητες της ΑΣΕΡ του Άσερ να ε, Έχει κυρίως από τους διαχειριστές διανομής πληροφορίες θα επιτρέψει μια καλή παρακολούθηση της αγοράς. Ο κύριος Χάνκελ είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι έχουμε πράγματι ε, μειώσει το θέμα αυτό στην πρότασή μας και θα ήταν δύσκολο να περιορίσουμε ακόμα περισσότερο το θέμα αυτό, διότι χρειαζόμαστε ένα όργανο, έναν φορέα συντονιστικό σε επίπεδο ρυθμιστικό. Και τέλος, νομίζω ότι με την βοήθεια αυτής της Επιτροπής, τον κύριο Τούρμερ προσωπικά, έχουμε για πρώτη φορά αντιστρέψει ε, την σειρά ε, της επιλογής. Όταν ήμουν εδώ την τελευταία φορά, είπα ότι δεν θα το δεχτεί η Επιτροπή. Φέτος ελέγχθηκε πρώτα ο πρόεδρος και μετά ε, χρειάστηκε ο Άσερ να επικυρώσει. Αυτή τη φορά επιτύχαμε ο πρόεδρος του Άσερ να εκλεγεί πρώτος ε, με ανοιχτό και διαφανή τρόπο. Και του ΣΥΕΡ, ε, του Συμβούλου, ήρθε μετά. Δεν ξέρω αν πρόκειται για δημοκρατικές αποφάσεις. Και αν ο ΣΥΕΡ, το Συμβούλιο, ελέγχει τον ίδιο πρόεδρο με το Άσερ αν είναι δημοκρατικό. Ε, ο ΣΥΕΡ, το Συμβούλιο αυτό, είναι ένα ιδιωτικό σώμα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το κατακρίνουμε αυτό. Αυτό είναι σημαντικό. Θα πρέπει η εκλογή ε, στον Νέισερ να γίνεται πρώτα με την κανονική διαδικασία και μετά ε, του Συμβουλίου με την βοήθεια των μελών αυτής της Επιτροπής και της Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μπορώ να είμαι συντομότατος. Έχουμε χρονική πίεση και για αυτό το φάκελο και για τους υπόλοιπους σχετικούς φακέλους. Τώρα, η σειρά των τροπολογιών και η σειρά με την οποία εργαζόμαστε προφανώς θα πρέπει να δείξουμε ευελιξία στο πώς δουλεύουμε, στο με ποια σειρά εξετάζουμε τις τροπολογίες λοιπά. Θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά. Θα ήθελα να σταματήσω λιγάκι, να σταθώ λιγάκι στα θέματα του κυρίου Χένκελ. Στην ε, έκκλησή του να μην αποδυναμώσουμε την πρόταση και μειώσουμε την προστασία. Είναι σημαντικό να κρατήσουμε αυτή την ε, γραμμή πλεύσης σε ό,τι κάνουμε πάνω σε αυτό το φάκελο. Και τέλος, είναι σημαντικό να ακυρώσουμε κάποιες από τις λανθασμένες αντιλήψεις που υπάρχουν για αυτή την πρόταση. Θα πρέπει να τα έχουμε όλα αυτά υπόψη μας στους επόμενους μήνες. Η συζήτηση ήταν επικοδομητική νομίζω. Ε, παραμένω αισιόδοξο και ας ξεκινήσουμε μάλλον να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά ούτως ώστε να φτιάξουμε ένα σωστό φάκελο στο τέλος. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους. Επίσης, να σας υπενθυμίσω ότι πρέπει να ψηφίσουμε στις 11 Δεκεμβρίου και για αυτό το θέμα. Κατά πάσα πιθανότητα θα αρχίσουμε στις 7 το, το βράδυ. Δευτέρα, Στρασβούργου, κανονίστε τα εισιτήριά σας για να είσαστε στο Στρασβούργο στις 7 η ώρα στην αίθουσα συνεδρίασης. Δευτέρα. Στρασβούργο του Δεκεμβρίου. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι. Τελευταίο θέμα. Ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων στον τομέα τη ηλεκτρικής ενέργεια. 233, 233 τροπολογίες υποβλήθηκαν συνολικά. Πολλή δουλειά υπάρχει ακόμα πριν φτάσουμε σε συμβαστικές τροπολογίες. Το σχέδιο έκθεσης παρουσιάστηκε από τον κύριο Τζανονάτο στις 11 Ιουλίου. Συνάδελφε, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως είναι προφανές, ο στόχος σε αυτή την περίπτωση είναι να μειώσουμε τον κίνδυνο στην ηλεκτρική ενέργεια, τον ηλεκτρικό κίνδυνο. Να αντιμετωπίσουμε αρνητικά ε, περιστατικά με, με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα και αλληλεγγύη και να μειώσουμε και τον αριθμό των εγκαταστάσεων κυρίως παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, γιατί σε ένα ορθολογικό σύστημα ο αριθμός των μεγάλων εγκαταστάσεων μπορεί να μειωθεί εξασφαλίζοντας ασφάλεια και βελτιώντας μας την ασφάλεια. Όπως ε, υπενθυμίσατε, υπάρχουν παραπάνω από 200 ε, τροπολογίες παρουσιάζονται στην πρόταση. Αυτό σημαίνει ότι χοντρικά δεν υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες για να βρούμε κοινή λύση τελικά. Ε, και προκύπτουν και κάποιες γενικές τάσεις, θα έλεγα, με βάση στα πλαίσια της έκθεσης, του σχεδίου έκθεσης μάλλον. Είναι διαφορετική συζήτηση που αφορά τις τροπολογίες που έχουν να κάνουν με το επίπεδο φιλοδοξία τριών από τι τέσσερι προτάσει τη πρόταση Κομισιόν. Καταρχά, το δεσμευτικό χαρακτήρα των μέτρων, πρώτον, την αρχή τη αμοιβαία αρρωγή, αμοιβαία συνδρομή και επίση ε, τι γίνεται με τι ε, διασυνοριακές περιοχέ. Νομίζω ότι αν ακούμε ένα τον άλλον, ε, θα μειώσουμε τις αμφιβολίες και θα μειώσουμε και τις αποστάσεις που μας χωρίσουν. Λοιπόν, καταρχάς για το θέμα των δεσμευτικών μέτρων. Νομίζω ότι είναι εκ των όνου κάνευ. Πάνω σε αυτό εδράζεται μεγάλο κομμάτι της συνολικής πρότασης. Δεν είναι δυνατόν να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια στον, ηλεκτρικό, στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς να βάλουμε κριτήρια μεγάλης διαλειτουργικότητας για την αξιολόγηση των επιδόσεων των εθνικών ε, συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Προφανώς η ενεργειακή ασφάλεια είναι κοινή ευθύνη των εθνικών κρατών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στα πλαίσια της αξιολόγησης των εθνικών επιδόσεων, η Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να παίξει πλήρως το ρόλο που της δίδουν οι συνθήκες. Ε, πάνω σε αυτό το σημείο υπάρχουν τροπολογίες και εδώ γενικά υπάρχει μεγάλη στήριξη για αυτό το στόχο, δηλαδή ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι δεσμευτικά. Αμοιβαία συνδρομή. Δεύτερο στοιχείο. Η τελευταία ενεργειακή κρίση του Ιανουαρίου του 2017 στην νότιο-ανατολική Ευρώπη μιλά από μόνη της. Όταν υψώνονται εθνικά ενεργειακά σύνορα, επιδεινώνεται η κρίση και η επίπτωση στα όμορα ενεργειακά συστήματα ε, είναι πολύ πιο σοβαρά. Ε, οι επιπτώσεις. Ε, κοινωνικά προβλήματα, οικονομικά προβλήματα κτλ. Επίση υπάρχουν υπηρεσίες, ε, συνδρομής, δημόσια ασφάλεια, προβλήματα που γεννώνται. Οι τροπολογίε για αυτό το σημείο κινούνται προς την κατεύθυνση και το πνεύμα της, του σχεδίου έκθεσης. Υπάρχουν κάποιες διαφορές για την εφαρμοσιμότητα σε ορισμένες προϋποθέσεις των μέτρων που δεν έχουν να κάνουν με την αγορά και που επιτρέπουν να επανέλθουν τα ενεργειακά σύνορα κάποιες φορές. Αλλά νομίζω ότι με βάση κάποιες τροπολογίες ότι η εφαρμοσιμότητα αυτών των μέτρων που δεν είναι της αγοράς θα πρέπει να επιτραπεί μόνο κατ' εξαίρεση. Ή θα πρέπει να επιτραπεί με βάση, ε, διαπιστωμένων, επί τη βάση διαπιστωμένων κριτηρίων. Και όταν η βοήθεια δίδεται θα πρέπει εν συνεχεία να αποζημιώνεται όπως πρέπει. Με βαση ε διαπιστωμενων διαπιστωμενων κριτηριων και οταν η βοηθεια διδεται θα πρεπει εν συνεχεια να αποζημιωνεται οπως πρεπει με βαση ε, τρόπους που έχουν συμφωνήσει τα μέρη που εμπλέκονται. Τώρα, ε, οι φορείς των ε, διασυνοριακών ε, περιοχών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ε, είναι όμως και αρκετά επίμαχο. Μιλάμε για ένα θέμα που μας αφορά, ε, αλλά μόνο έμεσα σε σχέση με, την, ε, με το σχεδιασμό της αγοράς. Θα ήθελα να σας πω ότι στις επόμενες συνεδριάσεις θα μπορέσουν μαζί με τους συναδέλφους που είναι σκιώδεις εισηγητές να συζητήσουμε και πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα διαφόρων link, των, ε, των διαφόρων δεσμεύσεων, ε, την, το σχεδιασμό της αγοράς και δηλαδή με, τη σχέση με την έκθεση Κάριντς και τις απόψεις των σκιωδών ε, εισηγητών. Τώρα, για τα περιφερειακά κέντρα συντονισμού, τα ROCS, Βλέπω ότι υπάρχουν τρία σενάρια με βάση τις ε, ιδέε των ε, συναδέλφων. Καταρχάς, να αναγνωρίσουμε πλήρω το ρόλο και τη λειτουργία του. Το δεύτερο σενάριο, ε, να έχουμε ένα τεχνικό επιχειρησιακό κέντρο, υπό αυτή την έννοια να λειτουργούν τα ROCs, υπό πολιτική αιγίδα και να δημιουργηθούν μακροπεριφέρειες από αυτά τα κράτη-μέλη. Το τρίτο σενάριο είναι αφισβητή τη νομική ισχύ του ροκ ή την απορρίπτει το ροκ και θέλει το status quo. Εγώ θέλω να υποστηρίξουμε την πρώτη προσέγγιση που σας είπα. Και επί της ουσίας και επί της μεθόδου. Στην, επί της ουσίας για λόγους ε, με αυτού που υποστηρίζουν και την ιδέα της αμοιβαίας ε, συνδρομής. Τα ROCs, αυτά τα κέντρα, ε, μας επιτρέπουν ε, μία ε, σταδιακή περιφερειοποίηση ε, στις ε, αρμοδιότητες της Ένωσης των κρατών μελών και των περιφερειών και μας επιτρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη επιχειρησιακότητα και να ξεπεραστούν τα εθνικά ε, ε, ε, συγγνώμη, ενεργειακά σύνορα. Τώρα, για τη μέθοδο. Νομίζω ότι με βάση αυτές τις ιδέες και άλλες ιδέες καλύτερα είναι να έχουμε μακρές ή μάλλον καλές ε, είναι να, έχουμε, να κάνουμε τις μακρές διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και εμείς να είμαστε ενωμένοι, να έχουμε αραγές μέτωπο εδώ στο Κοινοβούλιο. Τώρα, για τις τροπολογίες, πολύ σύντομα. Υπάρχουμε, υπάρχουν κάποια κριτήρια εμπιστευτικότητα στη δημοσίευση των πληροφοριών σε ό,τι αφορά ε, τα σχέδια και την αξιολόγηση του κινδύνου. Επίση, ε, άλλο θέμα είναι η συμπερίληψη των stakeholders στην, ε, στον καθορισμό τη μεθοδολογία για την προετοιμασία, διαχείριση και αξιολόγηση των κινδύνων και για του μηχανισμού λήψη των αποφάσεων και τι αρμοδιότητε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ΑΣΕΡ, Εθνικέ Αρχέ κτλ. Και εδώ η σχέση ανάμεσα στο, στα διάφορα θέματα ε, και στους διάφορους φακέλους θα πρέπει να τους ξαναδούμε. Αλλά συνολικά νομίζω ότι μπορώ να σας πω ότι δεν βλέπω μεγάλες διαφορές απόψεων μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Και έχω βαθιά πεποίθηση ότι θα μπορούσαμε να κλείσουμε γρήγορα το θέμα αυτό. Μετά από μια πρώτη συνεδρίαση που έγινε σε τεχνικό επίπεδο και με μια δεύτερη πρόσφατη συνεδρίαση σε τεχνικό επίπεδο με την συμμετοχή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ξανασυναντηθούμε ε, την επόμενη Τρίτη με του κοιόδης συζητητέ. Ε, επιτάπητος αυτή τη στιγμή είναι ένας πρώτος συμβιβασμό που τον έχω υποβάλει στους ε, βουλευτές και στους ε, συμβούλους και επ' αυτής ε, καταθέτουν οι συνάδελφοι διάφορες απόψεις και προτάσεις. Τώρα, με βάση τα όσα θα ακούσω σήμερα, θα ετοιμάσω μία επικαιροποιημένη ε, εκδοχή των συμβιβασμών που οι συνάδελφοι θα λάβουν αμέσως μετά, ούτω ώστε να είναι έτοιμοι για την πρώτη συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών, την επόμενη ουσιαστικά, που θα γίνει την Τρίτη. Προφανώς θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τη συζήτηση στο Συμβούλιο, όπου το Συμβούλιο μιλάει για σύνεση κυρίως για τη δεσμευτική ισχύ της και χαρακτήρα τη πρόταση, αλλά όχι μόνο, υπάρχουν και άλλε αμφιβολίε. Επίση, θα πρέπει να παρακολουθούμε παράλληλα τι γίνεται στο Συμβούλιο. Από τη μία, τι θέση θα έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέναντι στο Συμβούλιο, έτσι, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα την τάση ε, και το που πηγαίνουν οι διαθεσμικές ε, διαπραγματεύσεις και από την άλλη θα πρέπει εμείς να έχουμε την καλύτερη δυνατή ενωπημένη θέση ούτω ώστε να είμαστε σε ισχυρή ε, θέση απέναντι στο Συμβούλιο. Και η δική μας, ας πούμε, συνέντευξη ήταν πλατιά. Νομίζω ότι αρκούν αυτά. Πρέπει να σταματήσω. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για την προσοχή, καθώς και για την ε, συνεισφορά που μέχρι τώρα μου έχουν δώσει. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σίτα. Ε, ευχαριστώ Φλάβιο και ήταν πραγματικά μεγάλη η, παρουσία αυτή, η παρουσίαση αυτή σήμερα το πρωί. Δεν ήθελα να σας διακόψω γιατί έχουμε και λίγο χρόνο, αλλά να το θυμάστε ότι μίλησα σε 8,5 λεπτά. 8,5 λεπτά. Ρεκόρ. Να περάσουμε στους επόμενους ομιλητές. Ευχαριστώ. Νίτερ Μάιρ από το ΕΛΚΟ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και πρέπει να σκεφτώ τι ρεκόρ θα σπάσω εγώ. Εν πάση περιπτώσει, να σα πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ. Ήρθα μόλι από τη συνάντηση, από τη συνεδρίαση Πάναμα, όπου έχουμε 1.400 τροπολογίε. Άρα τα πράγματα καταλαβαίνετε μα φαίνονται πολύ απλά εδώ πέρα που μιλάμε για λιγότερε από 300 τροπολογίε. Φυσικά δεν ε, έχει να κάνει μόνο με την ποσότητα αλλά και με την ποιότητα. Να ευχαριστήσω λοιπόν τον εισηγητή, όχι μόνο επειδή έσπασε το ρεκόρ στην εισαγωγική του ομιλία, αλλά επειδή ε, επέτυξε πάρα πολύ μεγάλο πνεύμα συνεργασία. Από ό,τι φαίνεται η έκθεση ετοιμότητα του από τι τροπολογίε, δηλαδή φαίνεται ότι αποτελεί το πιο βατό ζήτημα από το φάκελο αυτό της ενεργειακής μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλό λοιπόν είναι να παρουσιαστούν οι φιλοδοξίες ε, της ε, έκθεσης και να κοιτάξουμε πώς μπορεί να υπάρχει χαμηλότερο κόστος ό,τι αφορά την ετοιμότητα και για τους πολίτες αλλά και για τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τους στόχους της ομάδας μας, θα θέλαμε μεγαλύτερη επικέντρωση, σε μεγαλύτερη ασφάλεια και μεγαλύτερη προσέγγιση βάσει της αγοράς, γιατί η σωστή ετοιμότητα ποτέ δεν οδηγεί σε επιδόνηση της κατάστασης, επιδόνηση της κατάστασης. Χρειάζεται νέα νομοθεσία για να καταργηθούν τα εμπόδια και η στρέβλωση της αγοράς και να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια. Η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών θα ενισχυθεί σε περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να υπάρχει σωστή διάσταση μεταξύ κρατών σε ό,τι αφορά και τις τεχνοριακές ροές και τα εμπόδια αυτά εξακολουθούν να υφίστανται ακόμα και σε περιόδους κρίσης και έτσι οι πολίτες επιβαρύνονται με περιττό κόστος και οι επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να συμμετέχουν στις διάφορες φάσεις της κατάρτισης του σχεδίου ετοιμότητας, προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια στη διαδικασία. Να έχουμε όμως υπόψη ότι η νομοθεσία θα πρέπει να εξασφαλίσει την εμπιστευτικότητα ευαίσθητων δεδομένων, γιατί αυτό ασφαλώς αγγίζει το σχέλο της ασφάλειας. Κάτι άλλο. Θα χαρώ να συνεργαστώ με τους κοιόδης για τις ε, συμβαστικές τροπολογίες. Είμαστε νομίζω σε σωστό δρόμο και προσβλέπουμε στις συνεργασίες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος από το ECR, ο, ο συνάδελφος Φόξ. Ευχαριστώ. Η ομάδα μου ε, υποστηρίζει την πρόταση της ε, Κομισιόν και να αυξήσει την αντίσταση και την ανθεκτικότητα σε για να έχουμε ένα προβλέψιμο πλαίσιο. Πρέπει όμως να διευρύνουμε το όλο και να περιλάβουμε χώρες των οποίων οι τομήσα ηλεκτρισμού είναι εντεταγμένη με τους δικούς μας. Θα πρέπει να έχουμε τους εταίρους ενεργειακής κοινότητας και άλλες τρίτες χώρες τα διατάξει δεν πρέπει να είναι μέτρα αγοράς και να δίνουν βεβαιότητα σε όλους τους εταίρους ότι θα λάβουν αντιστάθμιση και να δούμε πότε έχουμε μηχανισμούς υποστήριξης. Βεβαίως οι τροπολογίες είναι, συνάδουν με τα μέτρα για το αέριο και θα πρέπει να κρατήσουμε βεβαίως απόρριτες τις ευαίσθητες πληροφορίες. Βλέπουμε στις ομάδες συντονισμού της ηλεκτρικής ενέργειας ενισχυμένη αρμοδιότητα. Έχουμε τα νέα ε, κέντρα, τα περιφερειακά, ε, τα οποία είναι επιχειρησιακά, αλλά καλύτερα είναι να είναι ε, συνεργασίας, γιατί αυτό αντανακλά καλύτερα το ρόλο τους. και αυτό που προτείνουν ορισμένοι άλλοι θα μπορούσε να προτείνει φορτίο μεγαλύτερο σε έναν φορτωμένο τομέα καταλαβαίνουμε τους πρωταγωνιστές σε επίπεδο τοπικό, περιφερειακό και εθνικό. Νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε καλή συμφωνία για αυτήν την έκθεση. Θα συνεργαστώ με τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές. Δύο λεπτά. Δύο λεπτά. Εκ μέρους της Άλντε, ο συνάδελφος Πίτερσεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λαμβάνω τον λόγο εκ μέρους ε, της Γινιάχου, η οποία είναι σκιώδη εισηγήτρια. Βεβαίως ε, χαίρεται για την, ε, τα, την, τις τροπολογίες, για την ετοιμότητα. Πολλές τροπολογίες περιλαμβάνουν σημαντικές διατάξεις που ενισχύουν την πρώτη Κομισιόν σχετικά με τον ρόλο και αρμοδιότητες των διαφόρων ενδιαφερομένων φορέων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας για να υπάρξει μία ε, ισορροπία ανάμεσα στη διαφάνεια των πληροφοριών και στο απόρριτο των ε, πληροφοριών αυτών. Βελτιώνεται επίσης ο χρονισμός των διαφόρων ε, σεναρίων και ε, βελτιώνεται η τιμότητα. Τονίζει στις τροπολογίες τη σημασία της συνεκτικότητας ανάμεσα στις δράσεις και τα προγράμματα, τα εθνικά, τοπικά, περιφερειακά. Βεβαίως η συνεκτικότητα είναι σημαντικό θέμα σε αυτόν το φάκελο, όπως σε όλο το ενεργειακό πακέτο θα πρέπει να υπάρχει συμβατότητα με την με, τον, ε, με τον, ε, το δίκτυο ε, σε περιπτώσεις εκτακτές κατεπίγουσας ανάγκης και συνεργασία με τη ROX ή δεν ξέρω πώς θα τα ονομάσουμε. Βεβαίως θα συνεργαστώ με τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές για το θέμα αυτό. Εκ μέρους της Ρεμπέκα Χάρμς, σκιώδης εισηγήτριας για τους Πρεσίνους, ο συνάδελφος Σκλέτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα ότι δεν μπόρεσε η σκιώδη συγγήτρια να έρθει να συμμετάσχει στη συζήτηση. Θα διαβάσω τη θέση της για την εισήγηση. Όταν έχουμε περιπτώσεις κρίσεων, ε, τα κράτη-μέλη δρούν μονομερός, ε, πράγμα που δεν έχει νόημα ε, όταν έχουμε διασύνδεση. Πώς ε, στην κρίση ε, στην νοτιοανατολική Ευρώπη στην αρχή του έτους. Ε, οι Βούλγαροι για 70 μέρες επέβαλαν περιορισμό εξαγωγών και αυτό είχε βεβαίως επιπτώσεις στις γειτονικές χώρες και υπονόμευσε την εμπιστοσύνη στην αγορά και η κρίση αυτή και επίσης για τις γεννήτριες της Βουλγαρίας υπήρχαν 37 εκατομμύρια επιπλέον. Βεβαίως το σύστημα αυτό αντιμετώπισης των κρίσεων πρέπει να αντιμετωπίζεται με μέτρα εξάντε και εξ post. Εξάντε δεν είναι υποχρεώσεις, άμα δεν είναι υποχρεώσεις δεν πρόκειται να λειτουργήσουν. Προτείνει τροπολογία σας στην πρόταση της Κομισιό για να βοηθηθούν τα κράτη-μέλη, παραδείγματος χάρη. Αντί να αφήνουμε τα κράτη-μέλη στα σκοτεινά, οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να δίνουν κοινέ κατευθυντήριε γραμμέ στα κράτη-μέλη για να πώ προλαμβάνονται και να αντιμετωπίζονται περιπτώσει κρίσεων με μέτρα της αγοράς και μέτρα που δεν αφορούν την αγορά με βάση τα προγράμματα που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν επίσης τα κράτη για την διαπραγμάτευση συμφωνιών σε περιφερειακό επίπεδο. Επίσης, να δίνεται η προτίμηση στην αγορά και όχι σε μέτρα που δεν αφορούν τα αγορά. Οι, οι κανόνες της αγοράς που δεν αφορούν την αγορά θα πρέπει μόνο να χρησιμοποιούνται όταν είναι δικαιολογημένα. Επίσης, τα μέτρα ex θα μπορούν να ελέγχουν τα μέτρα και να προσδιορίζουν ε, την χρησιμοποίηση των μέτρων αυτών που δεν αφορούν την αγορά. Βεβαίως, όλα τα θέματα του μείγματος του ενεργειακού δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν σε αυτό το φάκελο, αλλά θα πρέπει να βρούμε λύσεις για να καλυφθούν ανεπάρκειες διάφορες δυνατότητες. Σας ευχαριστώ, συνάδελφε. Ζήλου Άγκα, σκιώδες εισηγητής από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ. Για τον κίνδυνο στην, ε, στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας έχουμε προτείνει διτές ε, τροπολογίες προς δύο κατευθύνσεις κινούνται που είναι σημαντικές κατά την άποψή μας. Καταρχάς, συμφωνούμε με την ανάγκη και τη σημασία των να έχουμε σενάρια κρίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αφορούν όλη την Ευρώπη δηλαδή, όμως δεν πιστεύουμε ότι θα πρέπει να έχουμε δίκτυα ε, ενεργειακών επιχειρήσεων και αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να δημιουργήσουμε αυτά τα σχέδια, μέσω των δικτύων δηλαδή. Γιατί στην πραγματικότητα γίνονται και δικαστές και δικαζόμενοι αυτές οι εταιρείε τελικά. Όχι. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε οργανισμού πιο αντιπροσωπευτικού που εκπροσωπούν το ευρωπαϊκό συμφέρον. Και από αυτή την έννοια προτείνουμε το ΑΣΕΡ να είναι οι ε, υπηρεσίες δηλαδή ε, συνεργασίας των ρυθμιστικών αρχών να είναι οργανισμός ε, που θα παίζει αυτό το ρολόγο το οποίο δρά και ανεξάρτητα από τα συμφέροντα των επιχειρήσεων του, του κλάδου. Δεύτερον, ξέρουμε ότι οι κανόνες της αγοράς σε περισσότερες, σε περισσότερες περιπτώσεις δεν συμβαδίζουν με το πνεύμα αλληλεγγύης που θα πρέπει να πριτανεύσει σε αυτήν την περίπτωση των κρίσεων, ας πούμε. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να βγούμε από αυτό το δόγμα της αγοράς και να έχουμε κανόνες που να βασίζονται στην αμοιβαία συνεργασία των κρατών μελών. Ακριβώς γι' αυτό η δεύτερη γραμμή τροπολογιών που παρουσιάζουμε είναι ότι πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να αναστείλουμε τους κανόνες της αγοράς όταν ε, επιδεινώνεται τα πράγματα. Γιατί μπορεί σε αυτήν την περίπτωση με τους κανόνες της αγοράς η κατάσταση κατεπήγοντος, η κρίση που έχει δημιουργηθεί να επιδεινωθεί. Πιστεύουμε λοιπόν ότι είναι σημαντικό να διαφοροποιήσουμε αυτή τη φάση. Δηλαδή, οι κανόνες αγοράς ισχύουν γενικά και αναστέλλονται σε περίπτωση κρίσεων. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Ο αντιπρόεδρος μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κ. Κόχλητσεκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό. Προφανώς όταν κάποια κρατημέλη ξεκίνησαν το επωνομαζόμενο πρασίνισμα της ενέργειας, είδαμε να υπάρχουν τεράστιες δοκιμάνσεις, κυρίως ε, σε χώρες ε, που ήταν ε, στην οδό διαμετακόμισης μεταξύ Γερμανίας και άλλων χωρών. Πέρσι μπήκαν μεταρρυθμιστές, φανταστείτε, στα δίκτυα. Χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν μετασχηματιστέ ε, σε ό,τι αφορά την προστασία των δικτύων από υπερβολική ενέργεια. Όταν υπάρχει για παράδειγμα ε, πολύ αέρα στη Βόρεια Θάλασσα μετά τι ε, ώρε αχμή για την χρήση ηλεκτρική ενέργεια. Να το έχουμε υπόψη μα αυτό γιατί αφαίρεση των εμποδίων μπορεί να βοηθήσει αφενός την αγορά, αλλά από την άλλη μπορεί να οδηγήσει και σε blackout όπως το παρελθόν στην Ιταλία. Είναι λοιπόν θετικό το ότι η έκθεση έχει κατατεθεί και έχει καταρτιστεί. Όπως ε, είναι μπροστά μας αυτή τη στιγμή, οι 300 τροπολογίες νομίζω ότι θα έχουν καταρτιστεί και αυτές με σωστό τρόπο και έτσι θα μπορέσουμε στο μέλλον να αναλάβουμε δράση και μάλιστα με τέτοιο τρόπο προκειμένου να λάβουμε υπόψη να, πηγές ε, στις οποίες δεν υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη. Φωτοβολταϊκά, για παράδειγμα. Έχω και εγώ φωτοβολταϊκά στην στέγη μου. Πρέπει να υπάρχει μια πηγή backup α, που να αντιδρά άμεσα αν υπάρχει πτώση της παραγωγής για τις ανεμογεννήτριες, τώρα στην Κεντρική Ευρώπη, επίσης είναι εξαιρετικά ανασφαλής πηγή. Γιατί κατά ελάχιστο, μάλλον γιατί παράγουν ενέργεια το πολύ 30% του χρόνου και πάλι λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει σύστημα ενίσχυσης. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Τη στιγμή που θα ξεκινήσουμε την πράσινη διαμόρφωση της παραγωγής ενέργειας θα πρέπει να υπάρχει και ένα σύστημα εναλλακτικής ε, παραγωγής η Τσεχία λαμβάνει μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή. Είμαι βέβαιος ότι και η Γερμανία θα ακολουθήσει σε μεταπιταχρονικό στάδιο, γιατί δεν είναι ακόμα συνδεδεμένη η Ανατολική Δύση στη Γερμανία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, λέγει ο Πρόεδρος. Ο κ. Ρουμπίχ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η προετοιμασία για ετοιμότητα για κίνδυνου στον τομέα της ηλεκτρικού παίζει σημαντικό ρόλο. Ξέρουμε ότι οι κυβερνοεπιθέσεις και η κυβερνοασφάλεια, για παράδειγμα, είναι κάτι καθημερινό πλέον. Και ως εκ τούτου είχαμε και την έκθεση προηγουμένω για τις αρχές ρυθμιστικές, αρχές για την ενέργεια. Και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι η συνεργασία μεταξύ Acer και BEREC ή της ε, εσωτερικής ε, αγοράς για την ενέργεια και για την ασφάλεια του δικτύου και με την ενίσα, θα πρέπει να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα η οποία θα λειτουργεί από κοινού. Και σε ό,τι αφορά την ετοιμότητα για τον κίνδυνο, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει συνεργασία αυτών των τριών ε, υπηρεσιών και θα καταστεί αυτό όλο και πιο σημαντικό, ξέρετε, στο μέλλον. Θα μπορούσαμε ενδεχομένω στην Επιτροπή να σκεφτούμε το ενδεχόμενο μια ε, έκθεση πρωτοβουλία για την ε, ενδεχόμενη συνεργασία μεταξύ των ε, υπηρεσιών αυτών στον τομέα αρμοδιότητα τη ε, ήτρε ενδεχομένω να γίνει μια μελέτη ή, εν πάση περιπτώσει, να υπάρξει μια σχετική πρωτοβουλία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, λέει και πρόεδρο. Κάποιος άλλος συνάδελφος, παρακαλώ. Ναι, ο κ. Σονκελή. Εν συντομία, όλα τα θέματα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και σημειώνεται σωστή πρόοδο η οποία φυσικά γίνεται μετά από σκληρή δουλειά. Και εσείς, ε, κύριε Πρόεδρε, στο... στην θέση της Προεδρίας διοργανώνεται ακροάσεις και το καθεξής. Ε, να θίξω το τελευταίο αυτό θέμα το οποίο ανέφερε ο συναδελφός Πολ το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα πρέπει να το τονίσουμε, γιατί είμαστε όλοι υπέρ της Ενεργειακής Ένωσης και της μεγαλύτερης συνδεσιμότητας και όσο πιο τα υποστηρίζουμε όλα αυτά, όσο πιο συνδεδεμένοι είμαστε, τόσο πιο ευάλωτοι είμαστε, κυρίως από πλευρά πλευράς ασφάλεια. Η συνεργασία λοιπόν μεταξύ των υπηρεσιών θα είναι πραγματικά αναπόσπαστο στοιχείο της μελλοντικής μας στρατηγικής. Χρειαζόμαστε πιο πολύ εμπειρογνωμοσύνη, πιστεύω, για να δούμε το πώς θα πρέπει στο μέλλον να δράσουμε προκειμένου να διευκολύνουμε όντως την ε, σύνθεση και μεταξύ κρατών μελών και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά την ε, απειλή της κυβερνοασφάλειας, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να πάρουμε πιο πολύ στα σοβαρά. Να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τον κίνδυνο, γιατί όπως σας είπα, όσο πιο συνδεδεμένοι είμαστε από την άποψη, τόσο πιο ευάλωτοι είμαστε, γιατί μπορεί να προκληθεί μεγάλος όλαθρος και καταστροφή. Ευχαριστώ, ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος και Τώρα να σας πω ότι γνωρίζουμε το ασυνήθιστο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα σου, Σον. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποφύγουμε ενδεχόμενη κρίση στην χώρα σας στο μέλλον. Θα ήθελα, λέει ο Πρόεδρος, να καλωσορίσω, τους βλέπετε άλλωστε, και το πίσω μέρος του αίθουσα. Έχουμε πάρα πολλούς καλεσμένους σήμερα το πρωί. Έχω καλεσμένους της κυρίας Βέρνερ από την Βόρεια Έση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που καλέσατε παρατηρητές των εργασιών μας στην Επιτροπή Ήτρε. Καλωσορίσατε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βάλτε τα ακουστικά, μην διστάζετε. Τίποτα, δεν ακούτε. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα, όχι φυσικά. Μάλιστα. Πολύ ωραία λέει ο πρόεδρος. να. Ναι. ήταν πολύ αυτοί που ήταν πάροντες από την αρχή μέχρι το τέλος, αλλά έχουμε μαζί μας τον διευθυντή του κύριο Μπόρχαρτ στον οποίο και θα δώσω το λόγο εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο, Πρόεδρε. Συνολικά η Κομισιόν καλωσορίζει όλες τις τροπολογίες στο σχέδιο έκθεσης. Το σχέδιο έκθεσης από μόνο του είναι πολύ καλό κομμάτι νομοθετικό ε, για το σημαντικό αυτό θέμα. Εάν η Κομισιόν έκανε ό,τι ήθελε, είναι, θα έκανε ακριβώ αυτό που είπε ο κύριο Νίντεμάιερ. Δηλαδή, θα προσπαθούσαμε να διατηρήσουμε πολύ ψηλά τη φιλοδοξία. Γιατί νομίζω ότι το σχέδιο έκθεσης με τις πολυάριθμες ε, τροπολογίες που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση βελτιώνουν το επίπεδο φιλοδοξία για να μην πω το αυξάνουν. Και προς τα εκεί θα έπρεπε να κινηθούμε. Με μεγάλη χαρά ακούω λοιπόν που και βλέπω ότι οι περισσότερες παρεμβάσει υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Δεν θέλω να επαναλάβω τα πάντα τώρα. Νομίζω ότι ο εισηγητής, ο κύριος Τζανονάτο, έκανε μια θαυμάσια εισαγωγή και πραγματικά είχε νόημα να ακούσουμε την ε, παρέμβαση του για αυτά τα 8,5-9 λεφτά ας πούμε και επί της ουσίας στηρίζω αυτό που είπε γιατί περιέγραψε πάρα πολύ καλά τι παίζεται εδώ πέρα με αυτό το φάκελο. Δύο μικρές παρατηρήσεις έχω να κάνω. Φυσικά δεν θα σε εκπλήξει σε αυτό το πλαίσιο ότι η Κομισιόν δεν υποστηρίζει αυτά που είπε ο κύριος Θηλουάγα, ότι θα πρέπει δηλαδή να αναστείλουμε τα μέτρα της αγοράς, γιατί μια λειτουργική, λειτουργούσα, εύρυθμη αγορά με διασυνοριακές ροές στην τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας είναι απαραίτητη για να επιληθούν τα προβλήματα σε περίοδο κρίσης. Και δεν είναι τμήμα, η αγορά δεν είναι τμήμα της κρίσης, γιατί αν πάμε πολύ, σε, πολύ γρήγορα σε μέτρα που δεν είναι μέτρα αγορά τι θα είναι, εθνικά μέτρα, α πούμε, θα είναι απαγορεύσεις εξαγωγέ, ας πούμε. Έχουμε δει τέτοια πράγματα να γίνονται και αυτό αντιβαίνει στην αρχή τη αμοιβαία αρρωγής, αμοιβαία συνδρομής και αλληλεγγύης που για μένα είναι η πρώτη και ακρογωνιαία αρχή όταν μιλάμε για προετοιμασία για να αντιμετωπίσουμε κινδύνους και κρίσεις. Η αμοιβαία συνδρομή και η αλληλεγγύη, αυτά είναι που πρέπει να υπάρχουν και μέσω των μέτρων της αγοράς Μπορούμε να το πετύχουμε, όχι μέχρι τη αναστολή των μέτρων. Τέλο, κύριε Ρούμπικ. Και ο άλλο Ευρωβουλευτή εκεί. Καταλαβαίνω απόλυτα τι είπατε. Η κυβερνοασφάλεια είναι θεμελιώδη και η πρότασή σα είναι ευπρόσδεκτη. Σα υποστηρίζουμε να κάνετε μια έκθεση ίδια πρωτοβουλία πάνω σε αυτό το θέμα. Και εμεί θα συνεισφέρουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ το Διευθυντή για την παρέμβασή του. Σας δίνουμε και το αργυρό μετάλλιο. Ε, γιατί ο άλλος ομιλητής ε, μίλησε 8,5 λεφτά, αλλά εσείς 6,5 λεφτά κτλ. Τώρα, νομίζω ότι όλοι οι παρόντες μίλησαν. Όλοι οι προσκεκλημένοι μας βλέπω έχουν τώρα τα ακουστικά τους. Είσαστε επισκέπτες από την Βόρεια Έση, Έση και είσαστε ευπρόσδεκτοι εδώ, είσαστε προσκεκλημένοι της Μαρτίνα Βέμπερ. Άρχισα να μιλάω πολωνικά τώρα, από εκεί που μιλούσα αγγλικά, γιατί να σας δείξω ότι 28 γλώσσες μπορούμε να μιλάμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, καν... Πουθενά άλλο δεν γίνεται αυτό, σε, καμία, σε κανένα άλλο πλαίσιο. Ο κύριος Ρομπίχ, κύριε Πρόεδρε, να σας ενημερώσω ότι χτες ε, εκφράστηκε το, δημοσιεύτηκε μία ένα global trend ε, από τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου. Πρόκειται για ένα δίκτυ ανάλυσης των παγκοσμίων τάσεων και έτσι λοιπόν την ε, μελέτη αυτή την ε, συμπληρώσαμε πλέον και με ανάλυση το Twitter. Κοιτάμε σε παγκόσμιο επίπεδο τι διαβιβάζεται και στο Twitter και διαπιστώνουμε τεχνολογικές τάσεις. Για μας λοιπόν θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό Επιτροπή Τεχνολογίας. Το Global Trend να το μοιράσουμε, αν γίνεται, στα μέλη της Επιτροπής ε, την επόμενη φορά, γιατί πιστεύω ότι αποτελεί μια πολύ καλή βάση για τις εργασίες μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Να ολοκληρώσουμε όμως πρώτα τη συζήτηση με τον εισήγητη. Να δώσουμε το λόγο. Θα είμαι τηλεγραφικός. Σας ευχαριστώ για την ε, υπομονή που είχατε, που ανοιχτήκατε τα 8,5 λεφτά μου. Νομίζω ότι αυτό δείχνει και τη μεγάλη φιλία που έχει η πόλη μου, η Πάντοβα, με την Πολωνία. Ε, ε, επίσης έχετε χρησιμοποιήσει, χρησιμοποιούν πάρα πολύ το βιτέλο και επίσης ο, ο Κοτσανόσκι, ο μεγάλος Πολωνός ποιητής, έχει σπουδάσει στην Πάντοβα. Ε, νομίζω ότι είσαστε πολύ ανεκτικός μαζί μου, ίσως επειδή έχουμε αυτούς τους ειδικούς δεσμούς. Να είμαι πολύ γρήγορος. Άκουσα μεγάλη προσοχή και εκτίμησα τις παρεμβάσει ε, και την τελευταία παρέμβαση του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα τα πούμε την Τρίτη για να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Thank uh, Άδελφοι, Έχουμε την ψηφοφορία στις 7 το βράδυ την Δευτέρα στο Στρασβούργο, την, την τελευταία σύνοδο του έτους. Έχετε τίποτα στα διάφορα να προσθέσετε. Τίποτα στα διάφορα. Να, να στείλετε όλα τα φύλλα, τα έντυπα που ο συνάδελφος Πολ Ρούμπικ πρότεινε και Έχουμε την επόμενη συνεδρίαση στις 6 Νοεμβρίου στις 3 το απόγευμα μέχρι τις 6.30, όχι 2.30, 3 η ώρα. Α, πολύ καλά. Στις 3 η ώρα. Στις 3 η ώρα. Άλλαξε η ώρα έναρξης συνεδρίασης. Ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι ότι καλή.